Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι χαρά μου σήμερα να σας καλωσορίσω όλους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας καλωσορίζω στη διάσκεψη αυτή. Καλωσορίζω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Φον Ρόμπαϊ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να καλωσορίσω τον Σωσέ Μανουέλ Παρόζο, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σωσέ Μανουέλ, σε καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη μου χαρά. Να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μεϊμαράκη. Μαζί θα συμπροεδρεύσουμε στην σημερινή συνεδρίαση. Σας καλωσορίζω λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην ε, έναρξη της Ολομέλειας της ε, Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας. Πρώτη φορά συνοργανώνεται μαζί με τα ε, Εθνικά Κοινοβούλια, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση. Η διάσκεψη αυτή συνοργανώνεται λοιπόν ε, φέτος ε, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν ε, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε Μεϊμαράκη, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε σε προετοιμασία αυτής της διάσκεψης. Το πνεύμα στο οποίο ετοιμάστηκε αποδεικνύει ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και έχουμε θέσει έτσι τις βάσεις για τη συνέχιση μιας επικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η περσινή διάσκεψη αποτέλεσε νέα σελίδα στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτισμού. Ήταν η πρώτη ευκαιρία για τα Εθνικά και για τους ε, εθνικούς και τους ευρωβουλευτές να έχουν μια συνεκτική προσέγγιση στο Ευρωπαϊκό, ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις πολιτικές του. Είχαμε λοιπόν ε, συμμετέχοντες από 26 κράτη και χαίρομαι που φέτος πάνω από 150 βουλευτές συμμετέχουν. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα και οι δύο πλευρές στόχο έχουν να βελτιώσουν τη συνεργασία και να αυξήσουν το δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για, το συντονισμό πολιτικών. Μαζί θέλουμε να σκεφτούμε την εμβάθυνση της ε, νομισματικής ένωσης και μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και ήδη πέρσι σημειώσαμε αποφασιστική πρόοδο στην θεσμοποίηση τη συνεργασία ανάμεσα στα εθνικά και, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φέτο θα εμβαθύνουμε τη συνεργασία αυτή. Προσβλέπουμε λοιπόν σε τρεις μέρες κατά τις οποίες θα εμβαθύνουμε τις πολιτικές και θα διασφαλίσουμε μια, έναν ανοιχτό διάλογο και την ομιμοποίηση των δομών ε, πολιτικής. Και θέλουμε έτσι να ενισχύσουμε τον εσωτερικό διάλογο. Οι συναντήσεις αυτής της εβδομάδας στόχο έχουν να αυξήσουν την αμοιβαία κατανόηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, όμως θέλουμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή πολιτική αρένα όπου να μπορεί να ασκείται ο δημοκρατικός έλεγχος. Είναι προσωπική μου πεποίθηση ότι εμείς οι ευρωβουλευτές και οι εθνικοί βουλευτές δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε εταίροι σε αυτής της προσπάθειας. Και είναι κοινό μας έργο να φροντίζουμε να λογοδοτεί η εκτελεστική εξουσία και να υπάρχει δημοκρατικό έλεγχο. Όλοι ξέρουμε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα λειτουργήσει μόνο εάν βασίζεται σε στενή συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, πραγματοποιεί ακριβώ, ε, μάλλον ε, λαμβάνει υπόψη της αυτή την πραγματικότητα. Έχει ενισχύσει τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τώρα μεγαλύτερη αναγνώριση και ευρύτερε εξουσίε στι πολιτικέ τη Ευρώπη, ιδιαίτερα όσον αφορά την επικουρικότητα, την ενημέρωση και τη συμμετοχή. Επιπλέον, η συνθήκη αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς αυτούς, θεσπίζοντας την διακοινοβουλευτική συνεργασία και μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει αναλάβει κάποια βήματα που να δείχνουν την δέσμευσή του να διευρύνει την κοινοβουλευτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φαίνεται στο ψήφισμα που υιοθέτησε το 2009. Και ναι, τότε φαίνονταν ρόδινα τα πράγματα για τον κοινοβουλευτισμό στην Ευρώπη, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, ε, μας έδειξαν μια διαφορετική πραγματικότητα η Ευρώπη ε, σκοντάφτει από τη μία κρίση στην άλλη και οι αποφάσεις ε, των Συμβουλίων Κορυφής επηρεάζουν όλους τους Ευρωπαίους. Οι αποφάσεις αυτές ε, λαμβάνονται όλο και περισσότερο και κλεισμένων των θυρών από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Οι πολλές συναντήσεις κορυφής, η αιμονή με τις συναντήσεις αυτές των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, Είναι κάτι που έχω περιγράψει κατά καιρού ω μια σύγχρονη διάσκεψη τη Βιέννη. Έχει μειώσει αυτή η αιμονή τον ρόλο που παίζουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σε εποχή κρίση αυτό μπορούμε να το δεχτούμε κατ' εξαίρεση, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε η εξαίρεση να μην γίνει κανόνας. Κυρίες και κύριοι, υπό την πίεση της διαχείρισης ε, την κρίσεων, εάν τα κοινοβούλια περιθωριοποιηθούν χωρίς να το νιώθουν αυτό, χωρίς να το συνειδητοποιούν, εάν τα κοινοβούλια, όπως ακούμε συχνά εδώ στις Βρυξέλλες, θεωρηθούν ενοχλητικός παράγοντας ε, και οι εργασίες τους θεωρηθούν ε, σπατάλη χρόνου, Αυτό είναι πραγματικά μια ανησυχητική εξέλιξη στην οποία θα πρέπει να αντιταθούμε. Στην διαδικασία για την Τραπεζική Ένωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι υπάρχουν ε, μέρη του μηχανισμού ε, ε, επίλυσης των διαφορών όπου προσπερνούν το κοινοβούλιο και είναι φυσικό ένα κοινοβούλιο να αντιτάσσεται σε κάτι τέτοιο. Περισσότερη Ευρώπη με λιγότερο κοινοβουλευτισμό δεν θα υπάρ... είναι κάτι που δεν θα υπάρξει με εμά. Και θετικό στην κρίση είναι ότι ενδιαφερόμαστε όλο και περισσότερο για το τι συμβαίνει στις γειτονικές μας χώρες. Αυξάνεται λοιπόν η συνείδησή μας ότι στην Ευρώπη βρισκόμαστε όλοι στην ίδια θέση, στην ίδια κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ένα καλό μήνυμα που θα μας ε, φέρει πιο κοντά στην εθνική διακυβέρνηση είναι ο διάλογος ε, με τα εθνικά κοινοβούλια. Η βάση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη αποτελεί μια κοινή κοινοβουλευτική βάση. Και γι' αυτό η κοινοβουλευτική εβδομάδα των εθνικών και ευρωβουλευτών. Η, έκθεση, η ετήσια έκθεση προόδου και η σχετική γνωμοδότηση αποτελούν σημαντικό βήμα για την διαμόρφωση μιας νέας μορφής ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ο τρόπος που συνεργαζόμαστε κυρίες και κύριοι είναι κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, διότι αυτό που κάνουμε τώρα αποτελεί καινοτομία. Αποτελεί μια νέα διάσταση κοινοβουλευτική συνεργασίας, αλλά αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Και γι' αυτό κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεστε εδώ. 150 βουλευτέ. μεγάλος αριθμός προέδρων επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, μια σειρά προέδρων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι με αυτό που ξεκινήσαμε θα συνεχίσουμε με αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό και ελπίζω ότι έτσι θα δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου θα έχουμε τις 28 ε, ε, τελεστικές αρχές ε, των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημιουργούμε έτσι ένα πλαίσιο κοινοβουλευτισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία στη συζήτησή μας αυτή την εβδομάδα. Κύριε Μημαράκη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ευρωβουλευτές και βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, είμαι ιδιαίτερο ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε μια πολυαναμενόμενη θα έλεγα διάσκεψη η οποία ανοίγει και επίσημα το κοινοβουλευτικό σκέλος της ελληνικής προεδρίας την πρώτη από τις επτά προγραμματισμένες διασκέψεις της Βουλής των Ελλήνων. Η διάσκεψη για την οικονομική διακυβέρνηση λαμβάνει χώρα για δεύτερη φορά μετά από αυτή του Βίλνιους που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο επί Λιθουανικής Προεδρίας. Έχει δε ως στόχο την εντονότερη συμμετοχή και διαβούλευση των Εθνικών Κοινοβουλίων επιζητημάτων που έχουν να κάνουν με τους πρόσφατους μηχανισμούς οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης τους μηχανισμούς δηλαδή που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την κρίση, να καλύψει ανεπάρκειες του οικοδομήματος της ΩΝΕ και να προλαμβάνει στο εξή παρόμοιες οδυνηρές καταστάσεις σαν αυτές που ζήσαμε. Επευκαιρία θα ήθελα να συγχαρώ τους Λιθουανούς συναδέρφους για την επιτυχημένη προεδρία που ολοκλήρωσε η χώρα τους μετά το τέλος του 2013. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η διάσκεψη λαμβάνει η χώρα στι Βρυξέλλες στο κέντρο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδος. Αποδεικνύει δε ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωκοινοβουλίου μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να παράξει. Ιδιαίτερα δε αυτή την κρίσιμη σημερινή συγκυρία και αυτό το γεγονός πρέπει να στηριχθεί από όλους. Οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκονται ανάμεσά μας σήμερα εκπροσωπούν τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τους Ευρωπαίους πολίτες. Και θέλω να τονίσω την ε, ιδιαίτερη συμβολή σε αυτή την προσπάθεια του Προέδρου του κυρίου Σούλτς για να επιτευχθεί αυτό, αλλά και να συγχαρώ και τους Προέδρους των Εθνικών Κοινοβουλίων που θέσαμε τα ζητήματα αυτά, τα συζητήσαμε, συνεργαστήκαμε και καταφέραμε να έχουμε αυτή την επιτυχημένη συνεργασία. Γιατί αυτό συμβολίζει τη διακριτή μεν αλλά συμπληρωματική αποστολή των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου. Η αγαστή συνέργεια των οποίων καλείται να εξαλείψει το δημοκρατικό έλλειμμα που δυστυχώς παρατηρείται σήμερα στην Ευρώπη από πάρα πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Η έλευση του 2014 δεν σηματοδότησε μόνο μια νέα αρχή για αυτή τη συνεργασία, για αυτή τη συνέργεια αλλά και μια αρχή για ολόκληρη την Ευρώπη της οποίας η οικονομία φαίνεται να επιστρέφει με αργά αλλά σταθερά βήματα σε αναπτυξιακούς ρυθμούς έπειτα από 18 ολόκληρους μήνες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ο πληθωρισμός σύμφωνα με προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και τα πρώτα σημάδια εξισορρόπησης της οικονομίας είναι πλέον εμφανή. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ευρωζώνη θα παρουσιάσει οριακή αύξηση ενώ εγχώρια ζήτηση εξαγωγές και ανταγωνιστικότητα επίσης θα κινηθούν με θετικούς ρυθμούς. βέβαια η αποσταθεροποίηση που προκλήθηκε στο οικοδόμημα της ονε λόγω ορισμένων λανθασμένων πολιτικών των κρατών μελών έλλειψης αποτελεσματικής εποπτείας από τις ευρωπαϊκές αρχές αλλά και αναπαρκών ευρωπαϊκών μηχανισμών όπως αποδείχθηκε παρατείνει την αβεβαιότητα η οποία κυριαρχεί και σήμερα και μία από τις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ευρώπη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διότι το υψηλό συσσωρευμένο δημόσιο χρέος σε πολλές χώρες, ο κατακαιρματισμός των χρηματαγορών, η ανεργία που έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ ιδίως στους νέους ανθρώπους θα συνεχίσουν να αποτελούν μεγάλο βραχνά και να αντισταθμίζουν οποιαδήποτε ωφέλη μπορεί να προκύψουν από τους βελτιωμένους δημοσιονομικούς δείκτες ταυτόχρονα διευρύνεται το χάσμα ευρωπαϊκού νότου και βορρά με τη συνεχή μεταφορά κεφαλαίων αλλά και εργατικού δυναμικού από τον μεν στο δε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο αυτό και λίγο στη χώρα μου. Οι χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της Ελλάδας που αναδείχθηκαν με το ξέσπασμα της κρίσης ανάγκασαν τη χώρα να μπει σε πρόγραμμα προσαρμογής και να υλοποιήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σκληρές αλλά εκ των πραγμάτων αναγκαίες πολιτικές. Πρόκειται για μια δίχως προηγούμενο δημοσιονομική προσαρμογή, θα έλεγα τη μεγαλύτερη και ταχύτερη που έχει επιτευχθεί ποτέ από μέλος του ΟΣΑ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε κατά 13,4 ποσοστιαίες μονάδες επί του ΑΕΠ ενώ το πρωτογενές έλλειμμα κατά 10,8 μονάδες με εμφάνιση θετικού προσήμου στο τέλος του 2013. Στο μέτωπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε ανακεφαλαίωση του τραπεζικού συστήματος, σε αποκρατικοποίηση άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, μεγάλες τομές στη δημόσια δίκηση, στη δικαιοσύνη, την υγεία, την παιδεία, το ασφαλιστικό σύστημα, την αγορά εργασίας και τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Ενώ όμως οι πολιτικές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, τα δυσανάλογα υψηλό κοινωνικό-οικονομικό κόστος έθεσε σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία των συγκεκριμένων προγραμμάτων προσαρμογής. Το ΑΕΠ μειώθηκε περίπου κατά το 1 τέταρτον σε σύγκριση με το 2009 και η χώρα έμεινε σε υφησιακούς ρυθμούς για 6 συναπτά έτη. Η ανεργία αγγίζει σήμερα το 27% και στους νέους το 57% και το 1 τρίτο του πληθυσμού δυστυχώς βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της στόχιας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Με απλά λόγια, οι αλλαγές ήταν και είναι επώδυνες για τους πολίτες των χωρών που ακολουθούν το πρόγραμμα προσαρμογής. Το βιωτικό επίπεδο επλήγησε σημαντικό βαθμό. Ειδικά στην Ελλάδα, όπως όλοι διαπιστώνουν πλέον, υπήρξαν δραματικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών και οι θυσίες τους είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ανάλογη είναι και η κατάσταση και στις υπόλοιπες χώρες του Νότου με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να εντείνεται το ρεύμα του ευρωσκεπτικισμού. Ρεύμα που βρίσκει θειασότες και σε πολίτες των υπολείπων κρατών μελών που δεν βλέπουν με θετικό μάτι την αυξανόμενη εισφορά στο πλαίσιο της αρχής της αλληλεγγύης και της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Συνεπώς, τώρα είναι κρισιμότερη από ποτέ η διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας των εν λόγω προγραμμάτων. Η απλή διαβεβαίωση ότι τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται και αλληλοποιούνται με αξιόπιστο, νόμιμο και διαφανή τρόπο και με τη συμμετοχή όλων των νομιμοποιημένων αρχών δεν είναι αρκετή και δεν πείθει πλέον τους Ευρωπαίους πολίτες. Άλλωστε έχουν παρατηρηθεί και έχουν ομολογηθεί λάθη και στα συγκεκριμένα προγράμματα. Αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη η παραγωγή αποτελεσμάτων ορατών στο μέσο πολίτη και η δημιουργία συνθήκων με στόχο το κοινό όφελος της ευρωπαϊκής οικογένειας και την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οράματος. Η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι βασικό στόχος του ευρωπαϊκού οράματος και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη για το 2014 που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Νοέμβριο αναφέρει ως κύρια προτεραιότητα τη δημιουργία ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επίτευξη ανάκαμψης διαρκείας. Το κυριότερο όμως εμπόδιο για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη είναι η περιορισμένη ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης σημαντικό πρόβλημα είναι η περιοριστική δημοσιονομική εξυγίανση. Στον αντίποδα αυτών, σημαντικό βήμα για την προώθηση της ανάπτυξης είναι η ταχεία εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ενιαίος ενωτικό εποπτικός μηχανισμός έχει τεθεί σε εφαρμογή ενώ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε πρόσφατα και τα κύρια χαρακτηριστικά του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης. Τόσο αυτοί οι μηχανισμοί, όσο και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των καταθετών, θα σπάσουν το φαύλο κύκλο εξάρτησης τραπεζών και δημοσίου χρήματος και θα διαλύσουν τις όποιες ανησυχίες υπάρχουν για τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου στόχος των κρατών μελών και ηγεσιών είναι να υπάρξει αφενός ένας υγιής τραπεζικός κλάδος θωρακισμένος έναντι πιθανών κινδύνων και αφετέρου να καταστεί εφικτή η αύξηση χορήγησης δανείων και αυτό προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης της πραγματική οικονομίας διότι αν δεν επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας δεν θα επιτύχουμε το στόχο μας την αντιμετώπιση δηλαδή των προβλημάτων των ίδιων των πολιτών, την αντιμετώπιση της κρίσης που πλήττει την ευρωπαϊκή οικογένεια από τη σκοπιά όμως του απλού πολίτη, του ανθρώπου και όχι με την απλοϊκή θεώρηση των αριθμών. Γνωρίζουμε άλλωστε πως ο στόχος της ανάπτυξης δεν είναι αόριστος. Έχει ως βάση τον πολίτη έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του και του συνόλου των πολιτών των κρατών μελών και την άμβληση των ανισοτήτων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2013 ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε πλήρως το ευρωπαϊκό εξάμεινο και η εφαρμογή του κρίθηκε πετυχημένη. Αν και βεβαίως πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης οι συστάσεις που εκδόθηκαν για τα κράτη μέλη κρίθηκαν αρκετά ισορροπημένες και υπήρχε η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ υιοθέτησης ξεκάθαρων και μετρήσιμων στόχων και ελευθερίας κινήσεων από το κράτος μέλος ώστε να επιλέξει ποιο μείγμα πολιτικής θα ακολουθήσει. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες είναι ουσιώδους σημασίας και γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις συστάσεις που αφορούν. Σύμφωνα με την έκθεση για το μηχανισμό επαγρύπνησης το 2014 τα περισσότερα κράτη μέλη σημείωσαν πρόοδο όσον αφορά τη διάρθρωση των ανισορροπιών τους. Και στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνία. Είναι ενδεικτικό το γεγονός πως η εγχώρια ζήτηση σε αρκετές οικονομίες υποχωρεί λόγω της ανάγκης αύξησης της αποταμίευσης των οικοκυριών από την μια πλευρά αλλά και από την άλλη των μισθολογικών εξελίξεων καθώς και των πιέσεων που ασκούνται στις επιχειρήσεις για τη μείωση χρέους με άλλα λόγια δηλαδή πάλι η μείωση μισθών η υψηλή φορολόγηση και η απουσία ανάπτυξης πλήττουν την οικονομική δραστηριότητα. σε συνδυασμό μάλιστα με την ανεργία οδηγεί σε επιδείνωση πολλών κοινωνικών δικτών σε επιδείνωση της ποιότητας ζωής. φέτος η περίοδος αυτή συμπίπτει με τη χρονική περίοδο των ευρωεκλογών και έτσι η όλη διαδικασία θα αποτελέσει πρόκληση για την ελληνική προεδρία ώστε να κατορθώσει να την ολοκληρώσει με επιτυχία και εντό των χρονικών περιθωρίων. Κλείνοντα θα ήθελα να τονίσω ότι ένα βασικό μάθημα που μα δίδαξε η κρίση είναι η ανάγκη για πολιτική εμβάθυνση πέραν τη οικονομική, δημοσιονομική και τραπεζική. Η πολιτική ολοκλήρωση είναι απαραίτητη ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ενισχυμένη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία στα επίπεδα που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο είναι κέρια σημασίας ο αποφασιστικός και ενεργός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η στενή του συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται οι αποφάσεις που παίρνονται να λαμβάνουν υπόψη την ευημερία της Ένωσης συνολικά, να αποτυπώνουν τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών έχοντας πάντα ως γνώμονα την εταιρική αλληλεγγύη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα τόσο σε κοινοτικό όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Δικαιοσύνη και διαφάνεια πρέπει να συνοδεύουν κάθε προσπάθεια, ούτω ώστε όχι μόνο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους, αλλά και η ευρεία αποδοχή τους. Τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα, αλλά και τις δύο επόμενες μέρες βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα και οι θέσεις που θα εκτεθούν εδώ θα είναι χωρίς αμφιβολία μεγάλου ενδιαφέροντος. Προσμένω λοιπόν σε ένα αγώνιμο και επικοδομητικό διάλογο. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω και να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική Προεδρία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μεμάρακη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του ε, Συμβουλίου, κύριε Προεδρέποντα, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σα ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να ε, μιλήσω κι εγώ στη διάσκεψή σα. Η εβδομάδα αυτή έχει, είναι πολύ σημαντική, ε, θα ακούσουμε πολλές φωνές και μέσα από τη συζήτηση Χρειαζόμαστε τις διαφορετικές επόψεις ε, για να θέσουμε τα δημοκρατικά θεμέλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι περισσότεροι εξημών έχουμε φιλόδοξα σχέδια για την Ευρώπη. Υπάρχει ένα ανεξάντλητο δυναμικό που μπορούμε ακόμα να εκμεταλλευτούμε και πρέπει να αναζητήσουμε το βέλτιστο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να το εκμεταλλευτούμε, έτσι ώστε η Ευρώπη να ανακτήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Γνωρίζω ότι μερικές φορές η φιλοδοξία αυτή οδηγεί σε ανυπομονησία και σε επικοδομητική κριτική, πράγμα το οποίο δεχόμαστε. Είναι όμως σημαντικό να μην ξεχνάμε από πού προερχόμαστε και πού βρισκόμαστε τώρα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, οι προκλήσεις αυτές ήταν μεγάλες και πριν την κρίση. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας επισημάνω πόσο δύσκολη ε, ήταν η κατάσταση έκτοτε. Η αλήθεια είναι ότι οφείλουμε να ανασχηματίσουμε, να επισκευάσουμε το σκάφος μεσούσης της κρίσης, της θύελας. Και το κάναμε αυτό. Η κρίση μας προσέδωσε την πολιτική δύναμη να προβούμε σε αλλαγές έτσι ώστε να είναι εφικτή η αλλαγή. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές ε, έμοιαζαν ασύλληπτες, αλλά με την πάρδο των ετών, βήμα προς βήμα, μπορέσαμε να αλλάξουμε το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που αναγνωρίζουν όλοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το τρέχον σύστημα είναι τέλειο, ότι έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας, ότι είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Κάθε άλλο, είμαι σίγουρος ότι η σημερινή συζήτηση θα αποδείξει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από σοβαρές συζητήσεις συμπεριλαμβανομένες και τη σημερινή. Αλλά αυτό θα δείξει εξάλλου ότι έχουμε κατορθώσει να προχωρήσουμε εντυπωσιακά πολύ σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, ενώ από τη μια οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρώπη, κυρίως στο στον τομέα της ανεργίας οφείλουμε να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης σε κάποια κράτη-μέλη, από την άλλη οφείλουμε να είμαστε και υπερήφανοι για τα βήματα που έχουν γίνει όσον αφορά την διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να θεωρούμε ότι δεν θα ξανασυμβούν αυτές οι τόσο κρίσιμες καταστάσεις και αν ξανασυμβούν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα-δύο χρόνια οι πολίτες ε, συζητούσαν τότε για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Και τώρα έχουμε εδώ την Ελλάδα παρούσα, προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόλις ακούσαμε από τον πρόεδρο του ε, ελληνικού κοινοβουλίου ότι η Ελλάδα νιώθει υπερήφανη που μπορεί να βρίσκεται στην προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πάμε στο θέμα των εξαγωγών. Μερικοί μίλαγαν για την κατάρρευση του ευρώ και τώρα τη βλέπουμε ένα νέο μέλος που προσχωρεί και αυτό στο ευρώ, τη Λετωνία, μετά από ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και μετά από ένα σκληρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο μόλις καιρό κάποιες κασάνδρες προέβλεπαν την κατάρρευση ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφατα προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλο ένα κράτος, η Κροατία και γίναμε 28. Ας μην ξεχνάμε ότι ορισμένε χώρες που βρίσκονται υπό επιτήρηση έχουν καλύτερες συνθήκες πλέον στις αγορές από άλλες χώρες που δεν ζήτησαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Και μάλιστα ορισμένες εξ σημείωσαν και μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης από πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα ορισμένε εξ βγαίνουν από το πρόγραμμα όπως το έκανε επιτυχώς η, Ιρλανδία, η Ισπανία όσον αφορά το πρόγραμμα τραπεζικής και οικονομικής βοήθειας ε, στο οποίο εντάχθηκε. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρισκόμασταν και πού είμαστε σήμερα. Να αναγνωρίσουμε ποιες ήταν ε, οι ελλείψεις από την αρχή. Σύντομα λοιπόν επιτρέψτε μου να σας ε, επισημάνω τις αδυναμίες με τις οποίες ήρθαμε αντιμετωπί κατά το προηγούμενο σύστημα. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνησης απέδειξε ότι ήταν πάρα πολύ ήπιο. Ήταν ανεπαρκές, ε, δεν ήταν δυνατόν να πιεστούν επαρκώς τα κρατη για να προβούν τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές. Μάλιστα μερικές φορές δεν ήταν καν δυνατό να ελέγξει κανείς ε, τους εθνικούς λογαριασμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αναγκασμένη να βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα που δεν ήταν πάντα τα σωστά, γιατί όλα αυτά συνετάσσονται κάτω από εθνική ευθύνη. Ε, έπρεπε λοιπόν να γίνουν μεταρρυθμίσεις στις ε, χώρες, αυτά όμως δεν γινόντουσαν αυτόματα και έτσι η Ευρώπη μπορούσε να τα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη, δεν μπορούσε όμως να παρεμβαίνει για τις απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές. Δεύτερον, σε επίπεδο δημοσιονομικό, ε, τα μέλη της Ευρωζώνης ε, με την προηγούμενη διακυβέρνηση είχαν καθορίσει στόχους, αυτούς τους στόχους τους ανέφεραν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν ήταν απόλυτα προσιλωμένα τα κράτη-μέλη στα προγράμματα αυτά. Και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι κάποια χρόνια πριν από την κρίση, πολλά, αν όχι τα περισσότερα κράτη της Ευρωζώνης, έσπαγαν, ξεπέρναγαν το δημοσιονομικό όριο που μόνοι τους είχαν ορίσει. Και η Κομισιόν ήταν εκείνη που έπρεπε να του υπενθυμίσει για την ανευθυνότητα αυτή, αλλά τότε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παραπάνω. Τώρα όμως είναι πλέον αποδεκτό ότι αν κάποια κρατημέλη δεν ξεπερνούν ή δεν ε, παραβιάζουν το σύμφωνο σταθερότητας, τότε αυτομάτως θα έρθουν αντιμέτωπα με ε, σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Τρίτον, δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ελέγξει κανείς ε, τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι εθνικές αρχές αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σε θέση να παρεμποδίσουν την μετακύληση των προβλημάτων. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομική επιτήρηση ήταν απόλυτα στα χέρια εθνικών αρχών και τι συνέβαινε σε κάποια τραπεζικά συστήματα, στα κράτη-μέλη, συνέβη το εξή οι εθνικές αρχές, οι εποπτικές αρχές δεν επισήμεναν καμία απολύτως δυσκολία. Και μόλις τώρα μπορέσαμε πλέον να εγκαθιδρύσουμε έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Ούτε υπήρχε ένα ευρωπαϊκό σύστημα για να επιβλέπει την εξυγένση και καθάριση των τραπεζών ακόμα και αν ήταν σαφές ότι μια χρεοκοπία μια τράπεζας ε, θα ήταν σχεδόν ανυπόφορη για μία και μόνο κυβέρνηση. Γιατί οι κυβερνήσεις και οι εθνικές αρχές, οι εποπτικές σε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, έδιναν τη δυνατότητα οι τράπεζες να σωρεύουν τα αποκαλούμενα επισφαλή δάνεια, τα οποία ξεπερνούσαν κατά πολύ το ΑΕΠ της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται υπό την ε, αρμοδιότητα, αν θέλετε, των εθνικών επιπτικών αρχών. Και επίσης, Όσον αφορά την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης υπήρχε ένα λάθος συνέστημα ασφάλειας. Υπήρχαν εποχές καλές, ε, τότε όμως ε, η κερδοσκοπία ξέφευγε από έλεγχο και κατόπιν ακολουθήσε η δύσκολη εποχή, η καιρή. Έτσι λοιπόν η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ε, πρόκειται να ολοκληρωθεί σε μία όμως ασταθή εποχή και μόνο προσπαθώντας να υπάρξει μία ουσιαστική εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης όπου ε, συντρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μόνο έτσι μπορέσαμε να δρομολογήσουμε έναν ικανό δρόμο για να διορθωθούν τα κακό κείμενα. Ας είμαστε λοιπόν απόλυτα σαφείς. Ενώ η κρίση δεν προκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα η κρίση δεν ε, ξεκίνησε καν εδώ, ήρθε εισαγωγή απ' έξω. Τελικά όμως η κρίση ήταν το αποτέλεσμα λανθασμένων και σε ορισμένε περιπτώσεις ανεύθυνων συμπεριφορών των χρηματοπιστωτικών αγορών και ε, λόγω της όρευσης εθνικών χρεών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια καθαρά δομικά δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και γι' αυτό ήταν αναγκασμένη να αντιδράσει μπροστά σε ιδιαίτερα δραματικές συνθήκες. Προσπαθήσαμε να είμαστε παράλληλα οι πυροσβέστες και εκείνοι οι οποίοι εκαλούντο να οικοδομήσουν ένα νέο οικοδόμημα για να ενταχθούν σε αυτό όλα τα κράτη-μέλη. Η κατάσταση βέβαια σήμερα είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε πιο σαφείς κανόνες, αυτό το οφείλουμε στο αποκαλούμενο εξαπλό πακέτο, το νομοθετικό πακέτο το οποίο ενέκριναν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Εστιάζουμε την προσοχή μας περισσότερο στον έλεγχο και έχουμε πλέον πολύ καλύτερο συντονισμό των εθνικών πολιτικών. Ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τώρα πλέον ε, είναι στοχευμένο και απόλυτα διαφανές. Έχουμε νέους κανονισμούς για τις τράπεζες, ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας και επίσης ε, πλέον ε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα ενοποιημένο σύστημα τραπεζών. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο μιας πραγματικής αμυγούς τραπεζικής ένωσης. Σε πολιτικό επίπεδο έχουμε αποδείξει επανειλημμένα ότι το ευρώ ήρθε για να μείνει, ότι είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, ότι έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας για να παραμείνει ε, το σκάφος αξιόπλο σε όλους τους ποταμούς και σε όλες τις συνθήκες. Η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά. Το αποτέλεσμα τώρα του αποτελέσματος δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τη δομή του συστήματος. Η επιτυχία βρίσκεται περισσότερο στο αποτέλεσμα, δηλαδή κρίνεται πλέον σε εθνικό επίπεδο. Βρίσκεται στη νόμιμοποίηση των προσπαθειών μεταρρυθμίσεων ε, σε κράτη-μέλη και στο σύνολο της Ευρώπης. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι από πλευράς αποτελεσματικότητας και νομιμοποίησης έχουμε τη λύση για όλα μας τα προβλήματα. Και οφείλουμε τώρα πια να κατανοήσουμε, όπως δεν συνέβη πριν από την κρίση, ότι αυτά που διαδραματίζονται σε μία χώρα πραγματικά μπορούν να έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες σε μία άλλη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε την οικονομική διακυβέρνηση, την κοινή και αυτό να το πράξουμε με έναν τρόπο που θα είμαστε δημοκρατικά υπόλογοι σε εθνικό αλλά και σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατόπιν τούτη, τούτου οι κανόνες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα. Αν δει κανεί λιγάκι τι θεσμικέ βελτιώσει που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια και την αναστροφή των χρηματοπιστωτικών εξελίξεων γιατί έχουν μειωθεί τα ελλείμματα. Διαπιστώνουμε ότι οι χώρες ε, που βρίσκονται σε πρόγραμμα όπως σας είπα τώρα πλέον ανακτούν τις δυνάμεις τους και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς ε, να αρνηθεί ότι έχει επιτευχθεί τεράστιο έργο. Βέβαια, οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνθήκες παραμένουν δύσκολε. και πάνω απ' όλα υπάρχει η τραγωδία αυτή της ανεργίας, κυρίως της ανεργίας των νέων. Γι' αυτό λοιπόν ε, στην έκθεσή μας για την ανάπτυξη του 2014 αναφέρουμε ότι αυτό που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να υπάρχει δημοσιονομική εξυγίανση με στόχο την ανάπτυξη, χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας γιατί ε, δεν θα πρέπει να επαλευθούν αυτά τα οποία έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν Επίσης, προάγουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές για την ανάπτυξη, για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία καμπή. Η ανάπτυξη επανέρχεται σιγά σιγά, έχουμε πλέον εισέλθει σε μια νέα φάση. Ε, βεβαίως δεν αρκεί το να ξεφύγουμε από την ύφεση για να πούμε ότι έχει ξεπεραστεί η κρίση. Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν δεν θα υπάρχει τόσο υψηλή ανεργία. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να συνεχίσουμε να στοχεύουμε στην ανάπτυξη και στην απασχόληση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ε, ε, ανάπτυξη, την ε, ανάκαμψη διαρκείας. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να υπάρχει πολιτική σιγουριά και σιγά σιγά να οικοδομήσουμε μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μερικές φορές ορισμένοι αναλυτές λένε ότι τα προβλήματα προέκυψαν λόγω του ότι η μία ή η αλλη απόφαση. Δεν είναι όμως αλήθεια αυτό και σας το λέω από την προσωπική μου εμπειρία. Όταν συζητάγαμε αυτά τα θέματα με τους εταίρους μας από την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Ρωσία, το ερώτημα που μας έκαναν ήταν δεν ε, ήταν ε, τι γίνεται με το έλλειμμα αυτής της χώρας ή το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μας έλεγαν τι θα γίνει τελικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το θέμα δηλαδή ήταν καθαρά πολιτικό. Κατόπιν τούτου όλα τα βήματα που έγιναν, γιατί έγιναν σημαντικά βήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παραδείγματος χάρη, αυτά μπόρεσαν να γίνουν διότι ο στόχος ήταν η εμβάθυνση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και επίσης, διότι τα κράτη-μέλη έδειξαν ότι είναι δεσμευμένα στο να μειώσουν το έλλειμμα και να προβούν σε μεταρρυθμίσεις. Ε, ξεκινήσαμε με την έκθεση που είχε παρουσιάσει ο πρόεδρος του Συμβουλίου από με μένα και με τον πρόεδρο του Eurogroup ε, και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μαζί είχαμε και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με όλα αυτά οι αγορές κατέληξαν συμπέρασμα ότι θα τα καταφέρουμε. Θα αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την Ευρώπη. Γιατί μερικές φορές ήμασταν και ο ασθενής του κόσμου. Ας πούμε στη συνδιάσκεψη των G20 ε, αυτό συνέβαινε. Όταν όμως ανακοινώσαμε τις αποφάσεις μας, τότε λοιπόν πολλοί συνειδητοποίησαν ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να υπάρξει η Τραπεζική Ένωση. Και δεν θα μπορεί να υπάρξει η Τραπεζική Ένωση πριν από τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης και καθάρισης. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι στο Κοινοβούλιο να επιτευχθεί συμβιβασμό πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και νομίζω ότι πρέπει να μετακινηθούν και τα δύο κόμματα. Δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα να λέει όχι εγώ δεν μετακινούμε καθόλου και οι δύο να το κάνουν. Και αυτό το στηρίζει ελληνική προεδρία και η Επιτροπή στηρίζει την ελληνική προεδρία για να προχωρήσει αυτή στην επίτευξη ω το δυνατόν στομότερα τη συμφωνία. Όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμότητα, το έχω πει επανειλημμένα ότι χρειαζόμαστε ένα πολυεπίπεδο σύστημα. Η λογοδοσία πρέπει να διασφαλίζεται στο επίπεδο εκείνο όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και βεβαίως να λαμβάνονται υπόψη και άλλα επίπεδα όπου θα προκύπτουν οι επιπτώσεις. Άρα δηλαδή, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και παράλληλα, εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είμαστε υπόλογοι απέναντι στο Κοινοβούλιο, είμαστε πρότιμοι να συνεργαστούμε συνεργαστούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια, βεβαίως στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αυτό ας πούμε το κάνουμε με το νέο σύστημα που υπάρχει, Δηλαδή, τον προηγούμενο Νοέμβρη για πρώτη φορά ε, δημοσιεύσαμε γνωμοδοτήσεις για σχέδια προϋπολογισμών. Πολιτικά έχουν υπάρξει εξελίξεις, έχουμε έρθει πιο κοντά και γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάλληλοι, θέλω να πω και το εξής. Πριν από κάποια χρόνια όταν οι πολίτες ρωτούσαν είναι καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωμοδοτεί για σχέδιο εθνικών προϋπολογισμών κάποιοι έλεγαν μα αν είναι δυνατόν. Σήμερα όμως λόγω της κρίσης αυτό συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα κράτη-μέλη ότι κάτι πρέπει να γίνει και είναι αυτονόητο ότι είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τα Εθνικά Κοινοβούλια διασφαλίζουν απολύτως τα δικαιώματά τους ε, στον προϋπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα βέτο ούτε να αλλάξει έναν εθνικό προϋπολογισμό. Όμως μπορούμε να συζητάμε και αυτό είναι σημαντικό γιατί με τον τρόπο αυτό θα εμβαθύνουμε την οικονομική διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, είναι καλύτερο και επίσης μέχρι τώρα υπήρχαν κάποια θέματα με τα οποία ασχολείται μόνο η πολιτική ελίτ ή κάποιοι εμπειρογνώμονες. Ακόμα δεν έχει ε, ριζωθεί σε δημοκρατικό επίπεδο ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι οφείλουμε να διαβουλευόμεθα με τους ε, εταίρους μας και ότι οφείλουμε να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουν όλοι αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ο τρόπος ε, με τον οποίο λειτουργούν οι χώρες ε, ε, οδηγεί στο να προκύπτουν επιπτώσεις και πέρα από τα στενά σύνορα ε, μιας χώρας. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία που διατρέχει αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεργαστεί περισσότερο και με το Ευρωπαϊκό και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι πλέον ξεφύγαμε από τα τεχνικά, ξεφεύγουμε και από τα θεσμικά, ας ε, ασχοληθούμε λοιπόν με το πολιτικό επίπεδο, την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχω πει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να συζητήσω με εσά τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να προσποιείται ότι ε, τα θέματα είναι τεχνοκρατικά. Όχι, όλα είναι δημοκρατικά και εκεί ε, διακυβεύεται το όλο παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο τον κύριο Μπαρόζο. Το λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος ο κύριος Βαν ε, Ρομπάη. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Βουλής, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόεδρε των Εθνικών μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, μέρη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Με ευχαρίστηση σήμερα είμαι εδώ μαζί σας αυτή την δεύτερη συνάντηση της διάσκεψης των Κοινοβουλίων δυνάμει του άρθρου 13 της Συνθήκης σταθερότητα. Διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις όπως η σημερινή είναι πολύ σημαντικές διότι βοηθούν τα κοινοβούλια που συμμετέχουν στο να ασκήσουν καλύτερα τον ρόλο ελέγχου που πρέπει να ασκήσουν σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας τους στην ε, ευρωπαϊκή λήψη αποφάσεων. Παρά το γεγονός ότι κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για την ε, οικονομική πολιτική της χώρας του και τον προπολογισμό της χώρας του, οι αρμοδιότητες αυτές τώρα ασκούνται σε ένα πλαίσιο μεγάλης αλληλεξάρτησης και γι' αυτό θα πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε αυτή την αλληλεξάρτηση. Η αλληλεξάρτηση βεβαίως είναι ιδιαίτερα στενή μεταξύ όλων αυτών που έχουν κοινωνόμισμα. Αλλά όπως αναφέρεται ρητά στη συνθήκη, στο άρθρο 121, έχει σχέση με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέγει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεωρήσουν τις οικονομικές πολιτικές τους ως ένα θέμα που τους αφορά όλους και να συντονιστούν με το Συμβούλιο. Κυρίες και κύριοι, η οικονομική κρίση η οποία μας έπληξε πριν από πέντε περίπου χρόνια ήταν η μεγαλύτερη πτωτική στροφή της οικονομίας του δυτικού κόσμου από την εποχή της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30 και απεκάλυψε τις ελλείψεις των εθνικών οικονομικών πολιτικές, πολιτικών της ε, ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς μας και της δομής της Ευρωζώνης. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέβαλαν υψηλό τίμημα για την έλλειψη εποπτείας των τραπεζών και για την ανεύθυνη διαχείριση κινδύνων του. Το χρέος του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ήταν μία άλλη από τις κύριες αιτίες της κρίσης και άλλα πολύ σημαντικά σφάλματα έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ευρωζώνη. Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας τα τελευταία χρόνια λοιπόν αναλώθηκε στην διόρθωση όλων αυτών των ελλείψεων και ανεπαρκειών. Έγιναν εξαιρετικές προσπάθειες και σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στις χώρες που πραγματικά ήταν στα πρωτοσέλιδα, αλλά όλοι μας χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε θέματα διαρθρωτικών αλλαγών και αλλαγέ μακροπρόθεσμε στην οικονομική μας κατάσταση. Εξετάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, βλέπουμε ότι ένα προφανές πρόβλημα και μια έλλειψη που είχαμε είναι ότι είχαμε, παρά το γεγονό ότι είχαμε μια κοινή χρηματοπιτωτική ε, αγορά, είχαμε πολύ λίγους κοινούς κανονισμούς και δεν μπορέσαμε να ρυθμίσουμε τα θέματα της εποπτείας της αγοράς. Ενεργήσαμε ο καθένας χωριστά και αναποτελεσματικά. Από τότε έχουν αλλάξει τα πράγματα, υιοθετήσαμε ένα σημαντικό ε, όγκο νομοθεσίας, ώστε να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε κοινού κανόνες, να ενισχύσουμε τους κοινούς μας για να μπορέσουμε τελικά να δημιουργήσουμε την ε, Τραπεζική Ένωση που θα είναι ένα σύστημα κοινή εποπτείας. Επίσης, είδαμε ότι οι κανόνες που αφορούν το χρέος και τα ελλείμματα δεν εφαρμόζονταν με τον κατάλληλο τρόπο. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε. Και τελικά μπορέσαμε να θεσπίσουμε διαδικασίες όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις ε, οικονομικές πολιτικές μεταξύ μας των κρατών μας. Τελικά, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, σε επίπεδο Ευρωζώνης, βλέπουμε ότι η συνθήκη του Μάστριχτ δεν προέβλεψε μία κρίση τέτοιας εμβέλειας και γι' αυτό θεσπίσαμε τους μηχανισμούς διάσωσης με αποκορύφωμα την Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και μπορέσαμε να συντονίσουμε καλύτερες τις οικονομικές μας πολιτικές έτσι όπως θεσπίζεται στη συνθήκη σταθερότητας. Συνεχίζουμε την εργασία μας με τη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης όπως αποκαλείται και κεντρική αρένα στην οποία διαδραματίζονται τα σημαντικά θέματα για την Τραπεζική Ένωση είναι το ΕΚΟΦΗΝ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ πιο λεπτομεριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν η αιστεία των περισσότερων συμφωνιών στις οποίες καταλήξαμε στο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του προηγούμενου μηνός. Το γενικότερο πλαίσιο αποτελείται από τρία μέλη από την εποπτεία, από την εξυγίανση και από την εγγύηση των καταθέσεων. Πρώτα απ' όλα εγγύηση των καταθέσεων. Υπάρχει νέα οδηγία που θα προβλέπει ένα ενοποιημένο σχήμα, έτσι όπως συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύο μέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεύτερον, στην εποπτεία. Ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας είναι κάτι το οποίο ε, τέθηκε σε εφαρμογή, ε, θα, με ένας μηχανισμός θα τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο με υπεύθυνη την κυρία Ντανιέλ Νουή. Και αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορα ε, τσεκ ε, της καλής υγείας στην οποία βρίσκονται οι τράπεζες. Τρίτο θέμα, η εξυγίανση. Η οδηγία για την ε, ανάπακαμψη και την εξυγίαση των τραπεζών που θα εναρμονίσει τους κανόνες τους σχετικούς συμφωνήθηκε επίσης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πιο σημαντικό από όλο είναι ότι οι Υπουργοί Οικονομικών μπόρεσαν να συνενέσουν για έναν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ως συμφωνία. Όλες αυτές η, η υλοποίηση όλων αυτών στους στόχος, η ταχύτητα με την οποία λήφθησαν αποφάσεις δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν. Για την Ευρωζώνη πρόκειται για το μεγαλύτερο άλμα που έγινε από την δημιουργία του ευρώ. Και αφήνουμε πίσω μας αυτό τον ε, αδύνατο κρίκο ή τον φαύλο σύνδεσμο που αφορά ε, τις προβληματικές τράπεζες και τα δημόσια οικονομικά. Επίσης, θα πω περαιτέρω ότι η Τραπεζική Ένωση ε, είναι η πλήρης δέσμευση όλων των ηγετών ώστε να δημιουργήσουμε μία ισχυρή και σταθερή ευρωζώνη. Η πολιτική μας βούληση παραμένει αταλάντευτη. Μέχρι το τέλος του έτους τα κύρια στοιχεία που θα συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσεις μας και στις εκθέσεις των τεσσάρων προέδρων, ώστε να έχουμε μία αυθεντική οικονομική και νομισματική ένωση, θα έχουν τελειοποιηθεί. Και ενώ βλέπουμε ποιες είναι οι ελλείψεις στην Ευρωζώνη, αρχίζουμε να κάνουμε μια νέα αρχιτεκτονική για την Ευρωζώνη, την οποία ανοίγουμε και σε κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Επίσης, επιτελέσαμε περαιτέρω πρόεδρο στο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για το, το... Ή, το οικονομικό, αν θέλετε, σκέλος της Οικονομικής Ένωσης. Η Οικονομική Ένωση, πέραν του ε, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του εξάπτικου πακέτου, του 6 pack, του 2-pack και του Δημοσιονομικού Συμφώνου είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και θέλουμε να το συμπληρώσουμε τώρα και με διάφορες εταιρικέ σχέσεις. Η ιδέα μας είναι να ενθαρρύνουμε τις βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες ώστε να, να μπορεί να λειτουργεί με υγιή τρόπο η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου επίσης επανήλθαμε στο θέμα της ε, ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, των θέσεων απασχόλησης. Κάναμε αποτίμηση του τι έχει γίνει μέχρι τώρα και της προόδου που αφορούν το σύμφωνο Ανάπτυξης και Θέσεων Απασχόλησης και με τον πρόεδρο Βέρνερ Χόιερ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων παρακολουθούμε τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ε, δανειοδότηση των οικονομιών μας και ιδιαίτερος για τον δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Νέα κοινοτικά κονδύλια για το 2014-2020 έχουν διατεθεί συμπεριλαμβανομένης και της πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και της πρωτοβουλία της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Έχει λοιπόν υλοποιήσει του στόχους της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα τελευταία έτος έχουμε κινητοποιήσει σε όλα τα δυνατά επίπεδα όλες τις δυνάμεις που μπορούμε για να μπορέσουμε να οθήσουμε την ανάπτυξή μας. Επιτρέψτε μου τώρα να επανέλθω στην σφαιρική εικόνα των σορευτικής εργασίας η οποία επιτελέστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βήμα προς βήμα, ώστε να μπορέσουμε να προσδώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα μέσα που χρειάζεται, ώστε πραγματικά να διαφοροποιηθούμε όσον αφορά την διαχείριση της οικονομικής μα. Ε, αλληλεξάρτησης. Πολλά πράγματα έγιναν βάσει των συνθήκων που προϋπήρχαν μέσω των ε, νομοθετικών διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλα θέματα απαιτούσαν τη δημιουργία νέων μέσων, τα οποία δεν διαθέταμε στο παρελθόν και τα οποία ήταν απαραίτητα να θέσουμε σε εφαρμογή μετά από έγκριση και κύρωση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Κάποια θέματα από αυτά αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, κάποια άλλα την Ευρωζώνη. Όλα βεβαίως τα θέματα έθεσαν το θέμα της ε, δημοκρατικής λογοδοσίας. Σε γενικά κανόνες η λογοδοσία για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο είναι βεβαίως κάτι το οποίο επιτελείται μέσω των εθνικών βουλών. Ενώ η λογοδοσία για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις εξασφαλίζεται από κοινού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν διπλή διασφάλιση, διτή νομιμότητα αλλά επίσης και διτή ε, πολυπλοκότητα στο θέμα αυτό. Όταν όμως μία απόφαση ενέχει και τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμη πιο πολύπλοκα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το είδαμε. Στο τέλος, τελικά, κάθε γραμμή λογοδοσίας βρίσκουμε ένα κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις διαφάνειας και αναγνωσιμότητας των διαδικασιών μας. Ένα κυρία θέμα το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι εθνικές βουλές μας είτε ελέγχουν μια εθνική απόφαση που λαμβάνει η κυβέρνησή τους ή την συμμετοχή της κυβέρνησης τους ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές αποφάσεις είναι σε θέση να διασφαλίσουν την λογοδοσία και έχουν τα απαραίτητα μέτρα για να το κάνουν. Το κύριο μέσο που διαθέτουν, η ικανότητα ελέγχου των ε, υπουργών τους σε κάθε περίπτωση, για κάθε κράτος μέλος, είναι να μπορέσει να οργανωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το δικό του σύνταγμα και την ε, κοινοβουλευτική του παράδοση. Σε ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί όλη αυτή η διαδικασία να διευκολυνθεί. Η θέσπιση διακοινοβουλευτικού διαλόγου, όπως αυτή της παρούσας ε, ε, συνδιάσκεψης, είναι επίσης ένα χρήσιμο μέσο. Όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις νέες αρχές στις οποίες έχουμε αναθέσει ειδικά καθήκοντα όπως ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας για τις τράπεζες και η αρχή εξυγίανσης που ενεργούν με κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές και πρέπει ό,τι κάνουν να γίνεται σε πνεύμα διαφάνειας και μηχανισμών αναφορά. Συμπληρωματικά θα πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει όπου χρειάζεται έναν ρόλο πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την, τον τα θέματα που αφορούν αυτούς τους νέους οργανισμούς. Αναμφίβολα μπορούν να γίνουν περισσότερα για να ενισχυθεί περισσότερο η δημοκρατική νομιμότητα και η λογοδοσία ε, στους μηχανισμούς που έχουμε θεσπίσει. Αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι οι προτάσεις ε, επί αυτού του θέματος θα πρέπει κυρίως να προέρχονται από εσάς, από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον τις ιδέες σας και τις υποδείξεις σας μετά από αυτή την διάσκεψη και από τα κοινοβούλια σας με τις ε, συνεχιζόμενους προβληματισμούς σας για τη θέσπιση της οικονομικής πολιτικής μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διαρθρώσουμε τη συζήτηση και δεν θα έχουμε το χρόνο να ακούσουμε όλους, ούτε θα έχει ο καθένας απεριόριστο χρόνο. Γι' αυτό προτείνω το εξής. Έχουμε 150 ομιλητές. Παρακαλώ να συμφωνήσουμε να περιορίσουμε το χρόνο ομιλίας σε δύο λεπτά. Δύο λεπτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ χρόνο ομιλία. Δεν ξέρω τι γίνεται στα δικά σα κοινοβούλια. Οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων έχουν συνήθω 4 με 5 λεπτά. Δύο λεπτά λοιπόν είναι αρκετά. Προτείνουμε λοιπόν να ακούσουμε κάθε φορά τέσσερις συναδέρφους από εθνικά κοινοβούλια και μετά έναν ευρωβουλευτή. Τέσσερα προς ένα. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε. με μια ε, διαδικασία την οποία θα σας εξηγήσω. Ακολουθούμε το πρωτόκολλο. Πρώτα θα ακούσουμε ε, τον Αντιπρόεδρο του ε, Ελληνικού Κοινοβουλίου, μετά από τα άλλα κοινοβούλια, μετά εκπρόσωπο του Γαλλικού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του Γερμανικού Bundestag και μετά έναν Ευρωβουλευτή, εφόσον ζητήσουν το λόγο. Μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει το λόγο κανένας ευρωβουλευτής. Το οποίο θεωρώ ότι είναι ε, μια χειρονομία ευγένεια απέναντι στους προσκεκλημένους μας. Ε, εάν συμφωνείτε λοιπόν, θα το κάνουμε ως εξής. Έχετε μπροστά σας ε, τις κάρτες σας για να ζητήσετε το λόγο. Σας παρακαλώ λοιπόν να δείχνετε την κάρτα σας αυτή. Θα τις μαζέψει κάποιος, Προτείνω λοιπόν να προεδρεύσω εγώ στον πρώτο γύρο. Στον δεύτερο θα προεδρεύσει ο συνάδελφος Μεϊμαράκης. Συμφωνείτε με τη διαδικασία αυτή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να σας πω επίσης ότι Μετράμε το χρόνο εδώ πέρα. Δεν είμαι πολύ δημοφιλή στο Ευρωκοινοβούλιο, ακριβώς επειδή σταματάω τους ομιλητές όταν ξεπερνούν το χρόνο ομιλίας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι αυστηρός. Ο κύριος Μεϊμαράκης ε, είναι γνωστός επειδή είναι διαφορετικός από μένα στο θέμα αυτό. Πρώτα λοιπόν ε, θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννη Τραγάκη. Παρακαλώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να ασχοληθώ με την Τραπεζική Ένωση κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, διότι αν αναλογιστούμε όλη η κρίση που ξέσπασε το 2008 ξεκίνησε ω χρηματοπιστωτική κρίση η οποία διαχύθηκε μετά και επηρέασε όλου του τομεί οικονομία. Είναι απόλυτα επιβεβλημένο η εμβάθυνση και ολοκλήρωση ΕΝΑ ξεκινήσει από τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία και την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάκτηση εμπιστοσύνη των αγορών και την ανάκαψη της πραγματικής οικονομίας στην Ευρώπη. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη διανυθεί με την απόφαση για την εφαρμογή του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Ενώ η ελληνική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να κλείσει και το θέμα του μηχανισμού εξυγίανσης μέσα στο εξάμεινο που διανύουμε. Έτσι ώστε ο οδικός χάρτης που προτείναμε, προτείνατε στην έκθεσή σας να γίνει πράξη όσο γίνεται πιο κοντά στα χρονικά όρια που εσείς θέσατε. Η εμπειρία ανέδειξε τους κινδύνους που ενέχει για όλο το οικοδόμημα της ΟΝΕ η μετακύληση του κόστους διάσωσης τραπεζών στους κρατικούς προϋπολογισμούς με άμεσο αποτέλεσμα τη διόγκωση του χρέους όπως είδαμε πρόσφατα και στην Κύπρο. Αντίθετα, είναι πολύ δικαιότερο να επομίζονται οι ίδιες οι τράπεζες τις αποτυχίες και τα λάθη των στελεχών τους, αντί να πέφτει το βάρος αυτό στις πλάτες των φορολογουμένων. Η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης είναι συνυφασμένη με ένα πιο σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα, πιο αποτελεσματική νομισματική ένωση. Ο συνδυασμός των δύο αυτών χαρακτηριστικών είναι ικανός να συμβάλλει στην πραγματική οικονομική σύγκληση και στην εξασφάλιση ρευστότητας που είναι απολύτω αναγκαία για να δώσει όθηση στην ανάπτυξη. Για το, για το σκοπό αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την επερχόμενη συνάντηση της ομάδας G20 το Φεβρουάριο του 2014 να είναι σε θέση να εκφράσει θετική της εμπειρία από το σχεδιασμό και την υλοποίηση τραπεζικής ενοποίησης, αναδεικνύοντας έτσι και την πρόσφατη πρόοδο στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτική σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Υιοθετώντα τη στάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδυναμώνει τη θέση τη στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, γεγονό το οποίο αποβάλλει τελικά, θα αποβεί τελικά προ όφελο των θεσμών και των πολιτών τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπερούτε Βισάιτε από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. κύριε Πρόεδροι, Συνάδελφοι από, το Εθνικό και τα από τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίε και κύριοι, καταρχά θέλω να ευχαριστήσω το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργάνωσαν την δεύτερη συνάντηση αυτή τη διάσκεψη. Όπω γνωρίζετε, η εναρκτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε ε, πέρσι τον Οκτώβριο στο Βίλνιου. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης στο Βίλνιους ελήφθησαν αρκετά σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την πρακτική οργάνωση των διασκέψεων αυτών αποφασίστηκε να ονομαστεί διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την ε, οικονομική για τη χρηματοοικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμφωνήσαμε να ξεκινήσει η διαδικασία του Βίλνιου για την προετοιμασία του τελικού σχεδίου των κανόνων και των διαδικασιών που θα οριστικοποιηθεί φέτος. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το όνομα της διάσκεψης και έτσι έχει στενέψει το πεδίο της. Επίσης δεν βλέπουμε να προβλέπεται χρόνος ε, για συζήτηση πάνω στον κανονισμό. Σε αντίθεση με την πρακτική της διακοινοβουλευτικής διάσκεψης, οι οργανωτές δεν έχουν προβλέψει επίσης την υιοθέτηση κάποιας τελικής διακήρυξης. Είμαστε πεπισμένοι ότι η διάσκεψη αυτή θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την ενδυνάμωση των εθνικών κοινοβουλίων ώστε να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των ε, χρηματοοικονομικών υποθέσεων. Και γι' αυτό θα θέλαμε να ανθαρρύνουμε τους ε, διοργανωτές αυτή και των επόμενων συναντήσεων να ε, να τηρήσουν τη συμφωνία που ελήφθη στο Βίλνιους που επιτέθη στο Βίλιο. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Κρίστοφ Καρέ από τη Γαλλία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την ε, συμπροεδρία την ελληνική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάγκη να εκδημοκρατήσουμε την όλη διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την σημασία της αγαστή συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να εμβαθύνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες έτσι όπως τι αρχίσαμε σήμερα και δυνάμε το άρθρο 13. Τώρα, θα ήθελα να πω το εξή: Θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ε, συμβιβαστική λύση στην οποία καταλήξαμε. Θα πρέπει να το κάνουμε. Εμείς ε, στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση θα συνεδριάσουμε στο τέλος του μηνός και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας και λαμβάνουμε υπόψη τι ακριβώς λέγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Νομίζω ότι την διαδικασία αυτή θα πρέπει να τη θέσουμε υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα όσον αφορά την ανάπτυξη. Δύο λόγια για να πω το εξής. Το 2014 Θα είναι αναμφίβολα έτος βελτιώσεων. Τα πράγματα εξελίσσονται αναμφίβολα θετικά, αλλά θα είναι κρίσιμη χρονιά παρόλα αυτά. Δεδομένου ότι θα πρέπει την ανάπτυξη να την συνοδεύσουμε με μέτρα, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ λεπτή. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Κυρίως την ε, εξισορρόπηση εξυγίανσης και ανάπτυξης. Ξέρω ότι οι προτάσεις επιτροπές έχουν ε, ε, αλλάξει και θα θέλω να επιμείνουμε περισσότερο στα θέματα του πολλαπλασιαστή και να το σκεφτεί και να το μελετήσει περαιτέρω το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μας. Ο κύριος Βαν Ρομπάι επίσης ανέφερε το θέμα του θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που βρίσκονται στο πρόγραμμα να Το λόγο λοιπόν έχει τώρα πρόεδρος του Bundestag ο κύριος Λαμάτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν ε, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σούλτς ε, και τον συνάδελφο κύριο Μεϊμαράκη για το ότι μας απίφθηναν αυτή την πρόσκληση από κοινού και με τον τρόπο αυτό κατέστησαν σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι αντίπαλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, είναι συνοδοιπόροι, είναι συνεταίροι, από κοινού επιθυμούν να αναλάβουν την ευθύνη. Βεβαίω, ε, αυτό που καθιστά όλη την υπόθεση δύσκολη αλλά και παράλληλα και πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ε, είναι το εξής, ότι δεν έχουμε τις ίδιες αρμοδιότητες, έχουμε διαφορετικές αρμοδιότητες. Άρα δηλαδή θα πρέπει να βρούμε κάποιο ευφυή τρόπο έτσι ώστε όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια να τα παρακολουθούμε κοινοβουλευτικά, να τα ελέγχουμε, να τα νομιμοποιούμε. Όπως ε, πολύ ωραία είπαν και ο κύριος Μπαρόζο και ο κύριος Βαν Χομπέι, ε, τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο έλαβαν χώρα πολλές και σημαντικές αλλαγές. Αλλαγές ε, οι οποίες ε, μας δίνουν πολλές περισσότερες δυνατότητες να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα τις κρίσεις και όμως αυτό να παρεμποδίζουμε να υπάρχουν κρίσεις. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το εύρος όλων αυτών των εργαλείων κατ' ουσίαν δείχνει ότι πρέπει να υπάρξουν αρμοδιότητες στον τομέα της Τραπεζικής Ένωσης, της δημοσιονομικής πολιτικής, ε, της ε, οικονομικής πολιτικής. Γι' αυτό κύριε Σούλτς, ε, αγαπητέ συνάλφε, αυτό που είπε συνάλφες από τη Λιτωνία το βρίσκω σωστό. Γιατί και εγώ τότε όταν είχαμε την πρώτη συνάντηση στο Vilnius και εγώ τότε είχα την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχουν και δικές μας αρμοδιότητες για τη δημοσιονομική αλλά και την μακροοικονομική πολιτική. Ε, αν δεν υπάρχει διάσταση απόψεων χρειαζόμαστε κατ' ουσίαν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνεργασίας ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα πλαίσιο το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ευέλικτοι. Βεβαίως δεν μπορούμε κάθε 14 μέρες να συναντιόμαστε και να συζητάμε. Γι' αυτό λοιπόν και αυτό το συζητήσαμε στη Λευκοσία, αν θυμάστε τότε. Είχαμε πει να ε, συνδυάσουμε τις αρμοδιότητές μας. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δουλέψουμε περαιτέρα. Και κάτι άλλο, όσον αφορά το συντονισμό, που είναι σημαντικός ο συντονισμός, ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη για απασχόληση δεν επέρχονται δια της επιφυτήσεως, ε, χρειάζονται οργάνωση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πολιτικά, ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποια είναι τα συμπεράσματά μας. Κατά την άποψή μου αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος αυτής της τακτικής κοινοβουλευτικής συνεργασίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάμερτ. Τώρα, το λόγο έχει εκ μέρους ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Επιπέδου, η συνάλφος Ιβάνα Μάριτετς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές και να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι σε τέτοιου είδους διασκέψεις συνειδητοποιούμε ότι για να επιτύχει το ευρωπαϊκό εξάμεινο χρειαζόμαστε πολιτική βούληση και πολιτική υποστήριξη. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο μας επιτρέπει να συνεδριάσουμε από κοινού και να μιλήσουμε για διάφορες σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που είναι διαφορετικές για κάθε χώρα μέλος αλλά η κοινή μας πείρα σε κάποια θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικού και είναι προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχουμε το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα του πολύ περιορισμένου επίπεδου εφαρμογής των συστάσεων της, Ευρωπαϊκού, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε όλοι μαζί ότι οι συστάσεις που γίνονται θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα κοινή προσπάθειας που καταβάλλεται από τις Εθνικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τα εθνικά προγράμματα θα πρέπει να συζητώνται πρώτα σε επίπεδο ε, κάθε εθνικής βολής, να επικυρώνονται και μετά να συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Ε, στρατηγική σημασία έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι προτεραιότητες και τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης θα πρέπει να συνδυάζονται με το στρατηγική σημασίας έγγραφο που αφορά την χρηματοδότηση όλων αυτών των πολιτικών. Θα πρέπει αυτά τα έγγραφα να διασυνδεθούν μεταξύ τους, ώστε να μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε σε μια θετική συνέργεια μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ την, τον κύριο Ροζάτη, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού από την Πολωνία. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του νέου συστήματο οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η προβλεπόμενη Τραπεζική Ένωση. Συμφωνώ ότι έχει σημειωθεί πολύ πρόοδο, ότι σημειώθηκε πολύ πρόοδο πέρσι, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει επιβραδύνει η πρόεδρο και θα ήθελα να καλέσω όλου του συμμετέχοντε σε αυτή τη σημαντική συζήτηση, ιδιαίτερα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, να πιέσουν τι εθνικέ κυβερνήσει του και του εκπροσώπου του ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή. Και θα ήθελα να αναφέρω δύο επιχειρήματα υπέρ της επιτάχυνσης της διαδικασίας. Το πρώτο επιχείρημα είναι οικονομικό. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές ε, ακόμα αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα. Υπάρχει ο φαύλος κύκλος ε, δημοσίου χρέους και τραπεζών που δεν έχει σπάσει ακόμα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα ε, στις νότιες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Και το άλλο επιχείρημα είναι καθαρά πολιτικό. Προχωράμε στις εκλογές και είναι πολύ πιθανό το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προκύψει μετά τις εκλογές να μην είναι τόσο διατεθειμένο να αναλάβει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες υπέρ της Ευρώπης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να ολοκληρώσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν το πολιτικό κομμάτι της Τραπεζική Ένωση πριν το τέλος αυτή τη θητείας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον ε, κύριο Χάρισον από το Ηνωμένο Βασίλειο, Πρόεδρο τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων Βουλή Λόρδων. Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο Παρόζο. Πιστεύει ότι τα χρήματα που έχουν διατεθεί στον μηχανισμό ε, εξυγίανσης, εάν αρκούν οι πόροι που έχουν διατεθεί. Και επίσης ε, πιστεύει ότι αρκεί διαβούλευση με 120 άτομα κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου για να λυθούν τα προβλήματα. Γιατί είπε ο πρόεδρος Βαρόσο ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ρόμπεϊ, διότι πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να το διατηρήσουμε. Και επίσης μπορεί να μας πει τι είδους συμβιβασμός θα πρέπει να επιτευχθεί για να διασφαλιστεί η επιτυχία του μηχανισμού εξυγίανσης και επίσης ο κύριος Ρόμπεϊ Συμφωνεί με αυτό που είπε ο κύριος Ροζάτη, ότι είναι απαραίτητο να κινηθούμε γρήγορα, να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Και τέλος, κύριε Σούλς, θα γνωρίζετε ότι η Βουλή των Λόρδων ολοκληρώνει την έρευνά της όχι μόνο πάνω στη δημοκρατικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πώς μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς, αλλά και πώς μπορούν τα Εθνικά Κοινοβούλια να προσθέσουν αξία σε αυτά που κάνετε εσείς, διασφαλίζοντας την δημοκρατική εποπτεία και εδώ στις Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο, αλλά και, στα, και στις 28 πρωτεύουσες. Να φροντίσουμε δηλαδή να υπάρχει επαρκή σε δημοκρατική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ τον κύριο Μπλαχά από τη Σλοβακία, πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ευχαριστώ <clears throat> Chcel by som že ľudia v Európe na Πρόεδρε, καταρχή, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ο κόσμος και στη Σλοβακία και αλλού θέλει κοινωνική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διαρριμένη σε 28 κράτη-μέλη. Είναι χωρισμένη σε πλούσιους και φτωχούς. Θα ήθελα να επισημάνω αυτό που είπε ο κύριος Σούλς και ο κύριος Μπαρόζο βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο σκάφο, βρισκόμαστε όλοι σε παρόμοια κατάσταση. Κάποιοι όμω ε, βρίσκονται πάνω στο κατάστρωμα, άλλοι βρίσκονται στο μηχανοστάσιο. Ε, και... μια ερώτηση προς τον κύριο Μπαρόζο. Υπάρχει κίνδυνος στον μηχανισμό εξυγίανσης ε, να υπάρχουν φορεί οι οποίοι θα αποκτήσουν περισσότερη εξουσία από τα κράτη-μέλη. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο δεν θα πρέπει να πέσει θύμα της παγκοσμιοποίησης. Ε, παρακαλώ τον... Ε, τώρα παρακαλώ τον κύριο Κιλκινέτα, βουλευτή από το Βέλγιο, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Merci, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Καλή επιτυχία στην Προεδρία και για όλες τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσετε στην Ελλάδα. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ κρατών ε, δεν μας βοήθησε. Θα πρέπει λοιπόν να συντονιστούμε. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε θέματα προϋπολογισμού έχουμε πρόβλημα τροχοπέδης που τίθεται στην ανάπτυξη της, της Ευρώπης. Και μπορούμε βεβαίως να δούμε ότι υπάρχουν ανομοιότητες στα θέματα πλούτου και ευημερία των κρατών μελών. Θα ήθελα να θέσω κάποια θέματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ασχοληθεί μαζί τους. Πρώτα απ' όλα, η κοινωνική και χρηματοπιστωτική συνοχή στις χώρες μας. Δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς καμία αντίδραση μπροστά στο κοινωνικό dumping που υπάρχει στις χώρες μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεύτερον, η αναζήτηση νέων οικονομικών πόρων, δηλαδή καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής και των ε, φορολογικών παραδείσων. Τρίτον, επενδύσεις στους τομείς του μέλλοντος, την έρευνα, στην ανάπτυξη, στους πράσινους τομείς και όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να αποτρέψουμε την επόμενη κρίση αντί να χρειαστεί εκ των υστέρων να πληρώσουμε τα σπασμένα και κυρίως να λάβουμε υπόψη τι θα γίνουν οι ΜΜΕ. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά τα θέματα να τα μελετήσουν, διότι αυτές είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία πιο υγιής, να έχει καλές επιδόσεις, να βοηθήσουμε τους νέους, διότι άκουσα τα θέματα της ανεργίας των νέων και για την Ελλάδα πόσο σοβαρά είναι. Παρακαλούμε λοιπόν ασχοληθείτε με όλα αυτά τα θέματα ε, τα οποία ανέφερα. Ευχαριστώ. Παπαδημούλη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Ευχαριστώ. Τα δύο λεπτά είναι λίγα για να πει κανεί τις απόψεις του. Θέλω να πω ότι δεν συμμερίζομαι το πνεύμα αυτοικανοποίησης και εξοραϊσμού που χαρακτήρισε τις ομιλίες των κυρίων Μπαρόζο, Ρομπάι αλλά και Σούλτς η ευρωπαϊκή οικονομία κινείται περί το μηδέν τα πηγαίνει χειρότερα από την αμερικανική οικονομία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με βάρβαρες πολιτικές λιτότητας σε πολλές χώρες έχει προβληματικό τραπεζικό σύστημα και ένα μεγάλο πρόβλημα χρέους. Θέλω να θέσω ορισμένα ερωτήματα και θα παρακαλούσα απαντήσεις προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Είσαστε ικανοποιημένοι από τις συνέπειες του προγράμματος που επιβάλλατε στην Ελλάδα προκαλώντας καταστροφική ύφεση, τεράστια ανεργία, εκρηκτικές ανισότητες, ανθρωπιστική κρίση. Γιατί βάλατε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην καρδιά της Ευρώπης. Προς τον κύριο Σούλτς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί χρειάστηκε να καθυστερήσετε τέσσερα χρόνια για να διαπιστώσετε ότι η Τρόικα στην Ελλάδα δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση και έλεγχο γιατί μέχρι τώρα αναβάλλεται όλοι μαζί μια ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα του χρέους. Γιατί το πρόβλημα του χρέους δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι και ευρωπαϊκό. Τι θα κάνετε για να ενισχυθούν οι πολιτικές συνοχής, περιφερειακής, εδαφικής και κοινωνικής μέσα στην Ευρώπη που έχουν αδυνατήσει τα τελευταία χρόνια στη διάρκεια της θητείας Μπαρόζο. Και τέλος, είναι δυνατόν όλα αυτά που λέει η συνθήκη της Λισαβόνας και οι ομιλίες σας να επιτευχθούν με ένα κοινοτικό προϋπολογισμό που είναι λιγότερο από 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αν η Ευρώπη δεν αλλάξει με το να στραφεί σε πολιτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της συνοχής θα συνεχίσει να μην αρέσει. Και γι' αυτό ευρωπαϊστές είναι αυτοί που αγωνίζονται για την αλλαγή στην Ευρώπη και για την ήττα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, επειδή ο κ. Ε, Παρόζο, ο πρόεδρος, ε, θα πρέπει και να αναχωρήσει γιατί έχει και άλλες υποχρεώσεις, θέλει να απαντήσει, να πάρει το λόγο. Yes, yes, of course. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά ε, στο μηχανισμό, στη διαδικασία, νομίζω πράγματι είναι τίμιο να αναγνωρίσουμε, όπως είπε και η φίλη μας από τη Λιθωνία και από τον Μπούνεσταγκο ο Λάμετ, ότι είναι η κατάσταση δύσκολη γιατί δεν ξεκινάμε όλοι από τις ίδιες προϋποθέσεις και απευθύνομαι σε εσά στα κοινοβούλια, σε εσά εναπόκειται να αποφασίσετε στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά από την εμπειρία που έκανα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, λόγω του κεντρικού ρόλου που είχαμε να διδαματίσουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να πω το εξή. Πρέπει να εξορθολογήσουμε, να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Γιατί πολλαπλασιάζοντας τις ευθύνες δεν διευκολύνει την κατάσταση. Και οποτεδήποτε συγκεντρώνει κανείς θεσμούς, δηλαδή ε, Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με 28 διαφορετικά εθνικά κοινοβουλία και μερικές φορές μιλάμε και για περισσότερα ακόμα, διότι ορισμένα ε, κράτη-μέλη έχουν όχι μόνο δύο κοινοβούλια, άνω και κάτω κοινοβούλιο, αλλά και πολλά περισσότερα περιφερειακά. Τα πράγματα λοιπόν δυσκολεύονται και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βελτιώνεται η διαφάνεια και η λογοδοσία. Να μην καταλήξουμε σε ένα δάσος, σε ένα οργανόγραμμα που κανείς δεν θα καταλαβαίνει τίποτα, όπου απλά θα έχουν πολλαπλασιαστεί οι ευθύνε και που τελικά θα έχουμε καταλήξει σε κάτι που είναι πολύ πιο περίπλοκο το οποίο δεν θα απλουστεύει τίποτα. Αυτό που τελικά ενδιαφέρουμε όλοι μας είναι η διαφάνεια, να είναι ευανάγνωστες, σαφείς οι αποφάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρώπης γενικότερα. Εμείς είμαστε ε, υπόλογοι απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή είναι η ουσία της ε, δημοκρατίας. Οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες απέναντι στα εθνικά κοινοβούλια. Άρα δηλαδή να υπάρχει συνεργασία σε διάφορα επίπεδα και όπως συμβαίνει μερικές φορές σε διάφορα θέματα, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο που τελικά να συμβάλλει σε αυτό που επιθυμούμε όλοι μας, που είναι το να είμαστε ελεγκτές να κυρίαρχοι της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μην προκύψει τελικά ένα μόρφωμα το οποίο θα περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα. Αυτό ήθελα να το πω οπωσδήποτε. Ε, υπήρξαν και άλλα δύο θέματα όπου έγινε, αναφέρθηκε το όνομά μου και κλήθη να απαντήσω. Το ένα αφορά την Τραπεζική Ένωση και το άλλο αφορά γενικότερα τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής. Όσον αφορά στην Τραπεζική Ένωση, και εδώ απευθύνομαι στην ερώτηση του συναδέλφου του κύριου από τη Βουλή των Λόρδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφής. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση η οποία δεν ήταν πιο ε, απλή από αυτή που τελικά συμφωνήθηκε. Παραδείγματος χάρη, όσον αφορά το θέμα της ευθύνης. Ποιος λαμβάνει την τελική απόφαση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που αποφασίστηκε τελικά και πάλι ήταν ιδιαίτερα περίπλοκο. Άρα δηλαδή η απάντηση προς εσάς. Και εδώ απευθύνομαι και στην παρατήρηση ε, του εκπροσώπου της ε, Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Εμείς θα προτιμούσαμε προφανώς να λαμβάνουμε τις αποφάσεις και να μην υπάρχει ένα είδος ε, συναέλευσης όπου θα συμμετέχουν δεν ξέρω πόσοι ε, επόπτες ή ε, ρυθμιστικές αρχές. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Υπήρξαν κάποιες ε, κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένης παρεμπιπτόνως και της Βρετανικής που ήταν η πιο άκαμπτοι σχετικά με το θέμα αυτό που δεν επιθυμούσαν πουδενή να έχει αυτές αρμόδιες η Επιτροπή. Δεν το ήθελαν. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε μια ομόφωνη απόφαση όλων των κρατών μελών όπου ε, μεκρίθη αυτό το συγκεκριμένο κείμενο που γνωρίζετε. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Δεν ήταν μόνο η Βρετανία, η Γερμανία, όχι σας το επισημαίνω. Ομόφωνη ήταν η απόφαση από όλες τις ε, κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλικής. Τώρα λοιπόν έχει προκύψει ένα πολιτικό πρόβλημα. Αν έρθει τώρα το Συμβούλιο με μια ομόφωνη απόφαση και το Κοινοβούλιο δεν συμφωνήσει με αυτή την ομόφωνη απόφαση και η διέστησή μου είναι επειδή έχω συζητήσει λιγάκι με τα ηγετικά στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι τελικά θα είναι μάλλον αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν δεν υπάρξει κάποια μετακίνηση προς την κατεύθυνση του συμβασμού. Εγώ λοιπόν και προς το Συμβούλιο και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέω να κατευθυντούμε προς τον συμβασμό. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, όπως είπε και κάποιος άλλος συμμετέχον κύριο σήμερα, το πρόβλημα ε, θα μετακυλιστεί στις αγορές. Και πραγματικά θα υποσκάψει τελικά τις εξελίξεις γιατί οι επενδυτές και οι αγορές ε, θα διαπιστώσουν ότι σε τελική ανάλυση δεν υπάρχει τραπεζική ένωση. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω αυτή την έκκληση. Ας δούμε τώρα ποιος θα είναι περίπου ο συμβασμός. Δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς αυτή τη στιγμή, γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει τίμια δουλειά και από τις δύο πλευρές. Όπως σας είπα, το Κοινοβούλιο, οι Κομισιόν θέλουν να συνεργαστούν, ο αρμόδιος επιτροπός μας θέλει να συνεργαστεί για να δούμε ποιε θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές ενός συμβασμού. Όμως, ας παραμείνει ανοιχτή η πόρτα για αυτή τη συμφωνία, γιατί αλλιώς ε, θα είναι ε, καταστροφή για όλους μας. Μία άλλη παρατήρηση που έγινε σχετικά με κάποια θέματα που δεν τα ανέφερα, παραδείγματο χάρη, α πούμε την εξασφάλιση των εγγύσεων. Μα δεν τον έφερα γιατί το θεώρησα δεδομένο. Αυτή ήταν ε, μια πρόταση επιτροπής, η διασφάλιση των καταθέσεων είναι προτάσεις της Επιτροπής. Έτσι λοιπόν είναι καλό που συμφώνησαν επ' αυτού και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αλλά ας δουλέψουμε τώρα σχετικά με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Τώρα όσον αφορά τη γενική πολιτική που ανέφερε νομίζω ο αξιότιμος εκπρόσωπος από τη Γαλλία. Ναι υπάρχει η στρατηγική 2020, ε, στρατηγική για την ανάπτυξη, ε, η ε, πράσινη, το πράσινο θεματολόγιο. Έχουμε καταθέσει πρόταση που όμως δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το Συμβούλιο. Ούτε το θέμα της ενισχυμένης συνεργασίας. Όλα δηλαδή αυτά τα θέματα που αναφέρεται σχετικά με την κοινωνική κατοχή, ε, κοινωνική συνοχή με και την αποφυγή του κοινωνικού dumping, η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και από αυτού συμφωνήσαμε. Γι' αυτό λοιπόν οι κυβερνήσεις ας προσπαθήσουν να αποφύγουν αυτό το κοινωνικό dumping που νομίζω είναι ε, αρνητικό για την Ευρώπη. Τελευταία ερώτηση που υποβλήθηκε από τον αξιότιμο ε, εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Έλληνα βουλευτή. Θα ήθελα να σε απαντήσω το εξή. Πρώτον, όσον αφορά το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, δεν ήταν δική μα η απόφαση. Τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ε, να συμπεριλάβουν το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στην Τρόικα. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτηση θα έπρεπε να τεθεί ω εξή. Να συνεχίσουμε με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Γιατί αυτό ήταν μια συνεκουανών προϋπόθεση για κάποιες κυβερνήσεις, απαρέγκλητος όρος δηλαδή, για να, ε, συμμετάσχει, να συμμετάσχει και το Διεθνές στο Ταμείο. Δεν ήταν πρόταση Επιτροπής. Ε, αυτή την ερώτηση μπορείτε να την κάνετε στις κυβερνήσεις, παρεμπιπτόντως γιατί όχι στην ελληνική, που το δέχτηκαν. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση τότε δεν μπορούσε να αρνηθεί, δεν είχε καμία δυνατότητα. Όσον αφορά το θέμα του προγράμματος και της δυσκολίας του προγράμματος, επιτρέψτε μου να είμαι ειλικρινή ειλικρινής απέναντί σας. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αν η Ελλάδα δεν εφάρμοζε το πρόγραμμα, σήμερα η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη. Εγώ είμαι πεπισμένος γι' αυτό και θέλω να πω στους Έλληνες φίλους το εξής. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις θυσίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Ελλάδα. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Αν η Ελλάδα δεν ήταν στην Ευρωζώνη ή αν δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θα έπρεπε να κάνει λίγο πολύ τα ίδια. Διότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν ήταν μόνο ένα δυσθεώρητο χρέος και προβλήματα στις τράπεζες, αλλά και διαρθρωτικά προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο ήταν θύμα, γιατί ήταν η πρώτη χώρα όπου όλα αυτά έγιναν ταυτόχρονα, σε αντίθεση με την Ιρλανδία. Και επιπρόσθετα από αυτές τις δυσκολίες η Ελλάδα αντιμετώπιζε και άλλες πολιτικής φύσεως δυσκολίες που δημιουργούσαν ανασφάλεια. Και οι αγορές θεωρούσαν ότι η Ελλάδα θα βγει από την Ευρωζώνη. Και τότε υπήρχαν και Έλληνες πολιτικοί που έλεγαν να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, από την ευρωζώνη. Και άλλοι το έλεγαν επίση, «Ε, αυτό δημιούργησε τεράστιε δυσκολίες. Όμω αυτό δεν έγινε. Στην Ιρλανδία, στην Ιρλανδία υπήρχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Γιατί λοιπόν το πρόγραμμα στην Ελλάδα ήταν τόσο πιο δύσκολο από ό,τι στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία. Διότι η Ελλάδα ήταν εκτέθηκε σε εσωτερικές πολιτικές δυσκολίες. Είχε να αντιμετωπίσει δύο ε, εκλογές, έγιναν κάποιες κουβέντες για να γίνει δημοψήφισμα και υπήρχαν και κάποιες εξωτερικές φωνές που δεν βοήθησαν τη χώρα. Έτσι λοιπόν, πέρα από τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές, όπως παραδείγματος χάνει το πολύ ψηλό επίπεδο φοροδιαφυγής στην Ελλάδα που είναι πολύ ψηλότερο από άλλες χώρες, όλα αυτά δημιούργησαν έλλειμμα εμπιστοσύνης. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, μπορούμε να συζητήσουμε εντάξει, αν το πρόβλημα ήταν τέλειο ή όχι. Προφανώς δεν ήταν τέλειο. Να είμαστε όμως και ειλικρινείς και ε, σχετικά με τις πληροφορίες που είχαμε τότε. Εμάς μας απασχολούσε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην καταστραφεί, να μην πτωχεύσει η Ελλάδα. Με αυτό το γνώμο να προχωρήσαμε. Και αν η Ελλάδα δεν ήταν στην Ευρωζώνη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν αναγκασμένη να πάρει χειρότερα μέτρα. Εγώ χαίρομαι που η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρωζώνη και χαίρομαι που εφέτος ε, η Ελλάδα ε, έχει να επιδείξει μικρή έστω αλλά κάποια ανάκαμψη. Αυτά είχα να σας πω. Δεν κάλυψα βέβαια όλες σας τις παρατηρήσεις αλλά προσπάθησα ειλικρινά να σας πω την δική μου την άποψη για όλα αυτά τα τόσο σημαντικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο τον κύριο Βαρόζο. Παρακαλώ την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την κυρία Άννη Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας καλωσορίζω και εγώ και εύχομαι και εξ ονόματος ε, των συναδέλφων κάθε επιτυχία στην ελληνική Προεδρία. Ε, ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο διότι το στίχημα θεωρώ ότι είναι ευρωπαϊκό τέσσερις μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Πρώτα απ' όλα στο σημείο που επισημάνθηκε ότι υπάρχουν ήδη τα πρώτα σημάδια της ε, ανάκαμψης της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας η οποία ωστόσο παραμένει εύθραυστη. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα και να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη δέσμευσή μας και στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική προσαρμογή. δεν φτάνει να το λέμε πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε κιόλας χωρίς διακρίσεις για να είμαστε ε, αξιόπιστοι απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες να το κάνουμε δηλαδή για όλες τις χώρες μέλη της ευρωζώνης όλες τις χώρες μέλη της ευρωπαϊκής ε, ένωσης και όχι μόνο όπως ε, επί του παρόντος προτείνει η ευρωπαϊκή επιτροπή για τα κράτη μέλη που έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο να το πράξουν. και το δεύτερο μιλώντας ε, ως ευρωβουλευτής ως αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου μιλώντας όμως ως κοινοβουλευτικός γιατί θεωρώ ότι ε, εκφράζω και του συναδέλφου από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια ε, το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω αφορά στο διακυβερνητισμό στην διακυβερνητική μέθοδο λήψης αποφάσεων. ο διακυβερνητισμός ήταν αναπόφευκτος ενδεχομένως ως ένα σημείο την πρώτη περίοδο της κρίσης που δεν είχαμε εργαλεία δεν είχαμε μηχανισμούς στη διάθεσή μας αλλά ο διακυβερνητισμός σήμερα όταν αναγορεύεται στην κυρίαρχη μέθοδο λήψης των αποφάσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο απειλεί την ίδια την συνοχή της ευρωπαϊκής ένωσης γιατί εκτρέφει τους εθνικούς εγωισμούς περιθωριοποιεί την κοινοτική μέθοδο που είναι η μοναδική μέθοδος λήψης αποφάσεων που διασφαλίζει τη θεσμική ισοτιμία ε, και την αποτελεσματικότητα στην προάσπιση του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος ως διαδικασία λήψης των αποφάσεων. θα ήθελα λοιπόν κύριε πρόεδρε κλείνοντας ε, να παρακαλέσω και εσάς ε, να παρακαλέσω την ελληνική προεδρία να υποστηρίξει με κάθε μέσο τη θέση αυτή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την επαναφορά στην κοινοτική μέθοδο στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων παντού και σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ τον κύριο Γκεργέρη, από, βουλευτή από το Εθνικό Κοινοβούλιο της Ιταλίας, από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Κύριος Γκεργέρη. Ε, παρακαλώ, ο κύριος ε, Γκάς από το Ηνωμένο Βασίλειο, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών... Ε, α, α, οκ. Okay. Yes. Uh, President Van Rompuy, uh, you stressed that the crisis... Κύριε Πρόεδρε Van Rompuy, Είπατε ότι η κρίση είναι και μια ευκαιρία να αναδιαστρωθεί η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Είπατε ότι έχουν ληφθεί θετικά βήματα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια. Πόσο μάλλον, αν σκεφτούμε, ότι έχουν γίνει πολύ τα πανηρές προσαρμογές στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχει γίνει έχουν γίνει αλλαγές στην Ευρώπη, αλλά τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν κατάρρευση στην εσωτερική ζήτηση και εσωτερική ε, υποτίμηση στα κράτη-μέλη αυτά. Το οποίο σημαίνει ότι το βάρος στην ε, Ευρωζώνη το φέρουν κυρίως τα κράτη της περιφέρειας. Οι μεγάλες χώρες είναι οι χώρες δανειστές και έχουν μεγάλο πλεόνασμα και έχουν συμβάλει σε περιορισμένο βαθμό στην εξέβρεση ισορροπίας στη ζώνη του ευρώ. Είναι αναποτελεσματική λοιπόν αυτή η προσπάθεια οικονομικά διότι έχει οδηγήσει σε αποπληθωρισμό στην ευρωπαϊκή ζώνη και έχει μειωθεί η εσωτερική ζήτηση στην Ευρώπη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, τι πιστεύετε ότι χρειάζεται στο εγγύς μέλλον από πλευράς της ε, οικονομικής διακυβέρνησης, ε, τι απαιτείται από την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική για να υπάρχει πιο συμμετρική προσαρμογή, ώστε να υποστηριχθεί η εσωτερική ευρωπαϊκή ζήτηση, που είναι πολύ σημαντική για να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, και πώς μπορούμε να έχουμε προσαρμογή στις ε, χώρες της περιφέρειας λιγότερο δαπανηρή από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν σημαντική τροποποίηση, χρειάζεται διαφορετική εφαρμογή των ε, μέσων ε, της οικονομικής διακυβέρνησης που έχουμε στη διάθεσή μας. Νομένο Βασίλειο, Πρόεδρο Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Uh, thank you, Mr. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κρίμα που έφυγε ο κύριος Παρόζο, διότι ήθελα να τον ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχει να κάνει με το σχέδιο που εκπονήθηκε πριν κάποιους μήνες, που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό αρμόδιο για το ευρώ. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι άκουσα τα όσα είπαν όλοι οι ομιλητές στο βήμα, αλλά δεν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Οι συνθήκες και η μέθοδος ε, νομοθεσίας στην Ευρώπη γεννά το ερώτημα ποιος κυβερνά την Ευρώπη και το ερώτημα περί δημοκρατικής νομιμότητας που εξετάζει η ΚΟΖΕΚ πολύ προσεκτικά και που είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κοιτάξτε τις δημοσκοπήσεις, κοιτάξτε το ευρωβαρόμετρο, κοιτάξτε τις διαμαρτυρίες για την ανεργία των νέων, κοιτάξτε το δημοκρατικό έλλειμμα. Τα εθνικά κοινοβούλια λαμβάνουν ε, την εξουσία τους από τις κοινοβουλευτικές εκλογές που είναι η βάση πάνω στην οποία ε, ε, λειτουργεί το Συμβούλιο των Υπουργών. Ακούω την Vivian Redding να λέει, για παράδειγμα, να έχουμε Ηνωμένε Πολιτείε ε, της Ευρώπης, να έχουμε περισσότερη πολιτική ένωση και ρωτώ τους ομιλητές στο βήμα, συμφωνείτε με την κυρία Ρέντινγκ. Όπως ρώτησα και τον κύριο Παρόζο πριν ένα χρόνο. Βρισκόμαστε τώρα σε θέση που άλλα μας λένε και άλλα λένε οι συνθήκες. Κανένας σε τούτη την αίθουσα δεν μπορεί να πιστεύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν απαραίτητο βαθμό νομιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν ε, την εξουσία που τους αξίζει. Οι συνθήκες θα πρέπει να αναθεωρηθούν ριζικά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ακούω την πολλοπλικότητα που περιγράφει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια λύση προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης. Τέλος, θα ήθελα να πω το εξής. Ε, θα ακολουθήσουμε την γαλλική ε, φράση ότι όσο περισσότερα αλλάζουν τόσο περισσότερα πράγματα παραμένουν τα ίδια ή θα έχουμε μια μεταρρύθμιση ώστε οι εθνικοί ψηφοφόροι να μπορούν να έχουν τον τελικό λόγο όσον αφορά το ποιο του κυβερνά. Παρακαλώ τον πρόεδρο τον κύριο Βανρομπάη να πάρει το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της ε, Βουλή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην ε, συζήτηση αυτή. Ήδη ο Πρόεδρος Μπαρόζο έχει απαντήσει τις περισσότερες ερωτήσεις που τέθηκαν στον πρώτο γύρο. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να δώσω κάποιες απαντήσεις στους άλλους ομιλητές. Πρώτα απ' όλα, εδώ αναφέρουμε την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, το τι κάναμε για την Δημοσιονομική Ένωση, για την Τραπεζική Ένωση. Όλα αυτά δεν είναι αυτοσκοπή. Ο απότερος σκοπός ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε την ε, αναδιάρθρωση, την ανασυγκρότηση της οικονομίας και να βοηθήσουμε την απασχόληση. Χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο από ό,τι ε, προβλέπαμε καταρχάς. Και βεβαίως χρειάστηκε να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες και να κάνουμε περισσότερες θυσίες. Αλλά αυτός είναι ο ίστατος σκοπός όλων των προσπαθειών που καταβάλουμε. Θα ήθελα να πω το εξής στους Έλληνες φίλους μας. Εγώ είμαι από μια χώρα η οποία στις αρχές του 80 είχε ε, δημόσιο χρέος 15% του έπτης. Στο ίδιο ύψος διαμορφωνόταν λοιπόν το δικό μας δημόσιο χρέος με αυτό των Ελλήνων σήμερα. Και χρειάστηκε να κάνουμε διόρθωση. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιήσαμε την υποτίμηση. Αυτό όμως δεν μας απέτρεψε από το να πάρουμε σκληρά και μη δημοφιλή μέτρα για να αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα, και τον, ε, ε, να εξισορροπήσουμε το όλο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Όλοι χρειάζεται να κάνουμε διορθώσεις όταν έχουν παρέλθει χρόνια, για να μην πω δεκαετίες, κακής οικονομικής διαχείρισης. Που, ποιος είναι ο στόχος λοιπόν των προσπαθειών μας. Αναθέρμανση της οικονομίας και της απασχόλησης. Η σταθερότητα είναι ένα μέσο, δεν είναι ένας αυτοσκοπός. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Και ο στόχος των οικονομικών μας πολιτικών είναι να αποκαταστήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατηρήση. Η δεύτερη αφορά τα δια, ε, κυβερνητικά και τα κοινοτικά μέτρα. Ακούστε, δεν θα κάνουμε τώρα μία συζήτηση ακαδημαϊκή από το τέλος, αλλά θα πω το εξής. Πρόκειται για μέτρα, δεδομένου ότι πάρα πολλές αποφάσεις λαμβάνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τα οποία μέσω της διακυβερνητικής διάστασης δώσαμε περισσότερη ενίσχυση, αν θέλετε, στην κοινότητα. Ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε τόσο πολλές αρμοδιότητες και την δύναμη να επηρεάσει την χρηματοπιστωτική πολιτική. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που έγινε ανευπροηγουμένου. Τώρα, υπάρχουν τα εργαλεία, τα μέσα που μας επιτρέπουν να διορθώσουμε τις ανισορροπίες χρηματοπιστωτικές, τις δημοσιονομικές και παρά το γεγονό ότι διαδραματίζει στον μηχανισμό εξυγίανσης και επίλυσης των κρίσεων η Κομισιόν, οι περισσότερες αρμοδιότητες είναι αυτές που έχουν τα κοινοτικά όργανα μεταξύ τους η μέθοδος μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά τελικά πού καταλήγουμε με όλα αυτά που κάνουμε. Προσπαθούμε με αυτή τη μέθοδο να ενισχύσουμε τον κοινοτικό ε, χαρακτήρα, αν θέλετε, το ότι κάνουμε. Θα ήθελα χωρίς να μακρηγορήσω να πω το εξής στους Έλληνες συναδέλφους. Εάν έχετε πάρα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος και ακόμη ε, ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όχι για ένα χρόνο, αλλά για πέντε διαδοχικά χρόνια, μία είναι η λύση. Να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε την ισορροπία. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο καθήκον, αλλά θα πρέπει να το αναλάβετε. Πολλές χώρες χρειάζεται να το κάνουν όταν έχουν ελλείμματα. Τώρα, ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν πλεόνασμα, αυτές που έλαβαν πριν να έρθει η κρίση τις, τα μέτρα και έκαναν τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές. Αλλά Επαναλαμβάνω, αυτό που ήταν κλειδί ήταν ότι έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα πριν να χρειαστεί να τα κάνουν. Γι' αυτό έχουν αυτό το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αυτοί όμως που έχουν πλεόνασμα εντός Ευρωζώνης διότι κάποιο μπορεί να έχει πλεόνασμα και εντό και εκτό Ευρωζώνη. Όποιοι είναι μέσα πρέπει να καταβάλουν περισσότερε προσπάθειε για να αποκαταστήσουν αυτή την ισορροπία, όπω είπα. Υπάρχουν χώρες που το κάνουν αυτό προσπαθώντας να αυξήσουν τον ε, ελάχιστο μισθό και υπάρχουν άλλες οι οποίες παρεμβαίνουν στον τομέα της παροχή υπηρεσιών. Και βεβαίω πρέπει να επαναλάβω, πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες και στις χώρες που έχουν πλεόνασμα, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι πριν από την εμφάνιση της κρίσης έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα, ενώ άλλοι δεν τα έλαβαν. Τώρα, η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης δεν είναι μόνο η δημοσιονομική εξυγίανση ή η αύξηση των μισθών. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Όταν αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη, αποκαθίσταται και το θέμα της ζήτησης. Και πότε γίνεται αυτό, όταν υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη επανέρχονται όταν όλοι βλέπουν ότι έχουν καταβληθεί οι σωστές προσπάθειες. Και μπορώ να σας δώσω παραδείγματα του πώς ο τα, διαφορετικά με συγχωρείτε, επιτόκια ε, καταδεικνύουν αυτό που λέγω. Θα σας δώσω το παράδειγμα της δικής μου χώρας. Κάποια χρονική στιγμή. Η διαφορά στα επιτόκια ήταν 350 μονάδες βάσης. Τώρα είναι 70 μόνο, διότι ελήφθησαν τα μέτρα με θάρρος, έγιναν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τους αντάμιψε για αυτό που έκαναν και το σύνολο των καταναλωτών και των αγορών που επανέκαμψαν. Και η αυξημένη απασχόληση. Μην υποτιμάτε λοιπόν όλα αυτό, αυτό το όλο θέμα της εμπιστοσύνης και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης που είναι και κάτι το οποίο αφορά γενικότερα την ε, οικονομία κάθε χώρας. Βεβαίως αυτό είναι μέρος της απάντησης. Η οικονομική εξυγίανση και η χρηματοπιστωτική ε, ε, εξυγίανση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι επίσης σημαντικές και όταν καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες μπορεί να είναι πιο ευέλικτη και η Κομισιόν στον τρόπο με τον οποίο βοηθά βραχυπρόθεσμα τις οικονομικές προσπάθειες που καταβάλλονται. Αλλά κάθε κράτος μέλος έχει την τελική ε, υλικό λόγο αν θέλετε. Ακόμη και αν ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση με πολύ αργότερους ρυθμούς από ό,τι περιμένουμε γιατί είναι πιο βαθιά από ό,τι υπολογίζαμε, πρέπει να υπολογίζουμε πάρα πολύ σωστά την διαρθρωτική ε, αλλαγή που θα κάνουμε ώστε να γίνει ισχυρή η οικονομία μας. Διότι με 1,5-2% δεν τα βγάζουμε πέρα. Χρειαζόμαστε περισσότερα Γι' αυτό οι μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές είναι πολύ σημαντικές και στις ε, χρηματαγορές και στην αγορά εργασίας. Και εάν είμαστε πιο ευέλικτοι σε θέματα ε, δημοσιονομικής ε, προσαρμογής, θα πρέπει να θεσπίσουμε περισσότερα μέτρα διαρθρωτικών αυτό ήθελα να σας τονίσω. Σας ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις και που κάνατε. Δυστυχώς θα πρέπει και εγώ να σας αφήσω. Αλλά πριν αποχωρήσω θα ήθελα και πάρει να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρεμβάσεις σας. Διότι έτσι ξέρουμε όλοι καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, κάτι άλλο που ξέχασα να πω για την ε, Τραπεζική Ένωση, γιατί είναι τόσο σημαντικό να καταλήξουμε τώρα στη συμφωνία. Αν δεν μπορέσουμε να βρούμε στα θέματα εξυγίανση συμφωνία που είναι τόσο σημαντικό για την Τραπεζική Ένωση, θα χάσουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Και μετά από τι ευρωεκλογέ η κατάσταση μπορεί να είναι περισσότερο πολλωμένη και θα μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλήξουμε συμφωνία. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω έκκληση στην ελληνική προεδρία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξέρω ότι υπάρχει πολύ καλή βούληση εκ μέρους όλων να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από το τέλος της παρούσης θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι διαφορετικά θα δείξουμε προς τα έξω ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ας μην δημιουργήσουμε λοιπόν αβεβαιότητα, Α καταλήξουμε σε μια συμφωνία Γι' αυτό το στοιχείο κλειδί για την σωστή λειτουργία της Νομισματικής και Οικονομικής Ένωσης και την επιτεύξη τη Τραπεζική Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο τον κύριο Βαν Ρομπάη. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η ώρα είναι, έχει περάσει ε, έξι το απόγευμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν το λόγο και να δώσω το λόγο στον κύριο Σούλτς για τα συμπεράσματα της σημερινής μας διάσκεψης, διαβεβαιώνοντας τον κύριο Ρομπάη ότι μέσα στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας είναι να υπάρξει συμφωνία στα θέματα που λέγαμε. Ο κύριος Σούλτς έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα πολύ σύντομα να μου επιτρέψετε να πω κάτι για την Τραπεζική Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρεται για συμβιβασμό. Βεβαίως ε, έχω την εντύπωση και μετά από όλα αυτά που άκουσα σήμερα ότι το Συμβούλιο δεν θέλει να μετακινηθεί ούτε ένα εκατοστό από τη θέση του. Ε, πώς θα γίνει συμβασμός. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και θέλω να σας πω ότι η απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ, του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών, όπως ελήφθη την τελευταία φορά, δεν θα συγκεντρώσει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως το ε, Κοινοβούλιο θέλει να ε, διαπραγματευτεί με το ΕΚΟΦΗΝ. Το ΕΚΟΦΗΝ βέβαια πρέπει κάτι να κάνει, να μετακινηθεί λίγο. Γιατί αυτό που μας είπατε σήμερα, το μήνυμα που λάβαμε, take it or leave it, μάλλον θα πάμε προς το leave δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα μετακινηθούμε ούτε εμείς. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος ε, Βαν Χομπέου, βεβαίως δεν είναι δικό του το Συμβούλιο, απλώς ε, προείσταται του ε, Συμβουλίου, θα πρέπει λοιπόν και εκείνος να κάνει κάτι για να μετακινηθεί το ΕΚΟΦΗΝ, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να βρούμε μια λύση. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις, κύριε Παπαδήμο, δεν ξέρω Πώς καταλήξατε στο συμπέρασμα, κύριε Παπαντιμούλη μάλλον να φέρει. Ε, εγώ επισκέφθηκα επανειλημμένα την Ελλάδα, κύριε Παπαντιμούλη, και έχω μιλήσει επανειλημμένα και με τον πρόεδρο του κόμματος. Νομίζω ότι είστε από το πρόεδρο του κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι δεν είναι. Ε, τρεις φορές διαπραγματευτήκαμε για το τι μπορούμε να κάνουμε για την βελτίωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Εγώ το έκανα αυτό, τρεις φορές το έκανα ω πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλλον κάτι δεν καταλάβατε καλά, κύριε Παπαντιμούλη. Εγώ ε, δεν ε, είπα αυτά που αφήσατε να Όσον αφορά την Τρόικα, αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Από ό,τι ξέρω, στις 29 Ιανουαρίου θα έρθουν οι συνάδελφοί μας στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε με τους συναδέλφους μας που παρόντος, παρεπιπτόντος είναι ε, παρόντες εδώ. Είναι ο κύριος Κάρας και ο κύριος Νόκα και μπορείτε αν θέλετε κατηδία να τα πείτε να πω κάτι για τον κύριο Κέσ. Κύριε Κέσ, αυτά που είπατε, αυτό το απόφευγμα δεν είναι γαλλικό. Είναι ένα απόφευγμα από το θαυμάσιο μυθιστόρημα Λεοπάρ του Τόμας Σιντι Λαμπεντούζα που λέει το απόφευγμα όλα πρέπει να αλλάξουν για να παραμείνουν όσα έχουν. Το θέμα είναι αν θέλουμε να παραμείνουν όσα έχουν γιατί έχω την εντύπωση ότι ε, πολλοί δεν θέλουν να παραμείνουν τα πράγματα όσα έχουν. Το θέμα είναι λοιπόν ε, τι ορίζουμε το ότι να μην όλες έχουν. Γιατί αν η ιδέα της ε, διεθνικής δημοκρατίας που εγώ θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης κατά τον 20ο αιώνα, αν θέλουμε να το σώσουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά. Αλλά τουλάχιστον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μπορώ να σας πω ότι αυτή η ιδέα της ε, διασυνοριακής, της διεθνικής δημοκρατίας δεν τίθεται σε συζήτηση επουδενή. Γιατί αν επρόκειτο να τεθεί στη συζήτηση θα προσέκρουε σε ότα μία κόντων. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη ε, συζήτηση για το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Πακέτου και την Προεδρία θα αναλάβει ο συνάδελφός μου ο κύριος Ότμαρ ε, Κάρας ε, που νομίζω ήδη κάπου εδώ βρίσκεται και του εύχομαι του κυρίου Κάρας ευόδοση των εργασιών. Επιτρέψτε μου εγώ να κλείσω το πρώτο τμήμα των εργασιών μας. ελπίζουμε ότι θα βγάλουμε τελείω νέο κείμενο μετά θα δούμε μεταξύ μα, Οπότε έχω βάλει εδώ Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, Παρακαλώ. Πώς είναι η γραμμένη πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή συνεδρίαση. Η διακοινοβουλευτική συνεργασία αποκτά σήμερα μια νέα διάσταση μέσω της συνδιοργάνωσης μιας πολυεπίπεδης διάσκεψης με την εμπλοκή διαφορετικών επιτροπών τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα εθνικά κοινοβούλια. Προσδοκούμε σε μια ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συνέβρεση στην οποία θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα και ρεαλιστικά ο παλμός της Ευρώπης ως συνόλου αλλά και της κάθε χώρας ξεχωριστά στο κρίσιμο ζήτημα της οικονομικής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την ε, ε, πραγματοποίηση και της τρέχουσας διάσκεψης και έχοντας αποκτήσει την εμπειρία της συνδιοργάνωσης θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε εκ νέου τη συζήτηση για τον κανονισμό λειτουργίας ετέθη το θέμα σύμφωνα με τον ακόλουθο οδικό χάρτη. Στις αρχές Φεβρουαρίου θα στείλουμε ξανά το σχέδιο κανονισμού της Λουθανικής Προεδρίας με ενταγμένες προτινόμενες προτάσεις μας με προθεσμία υποβολής νέων τροπολογιών ως τα μέσα Μαρτίου από τα εθνικά κοινοβούλια. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ως τα μέσα Απριλίου μια σύνθεση για ζητήματα που εκκρεμούν θα συζητηθούν πριν τη διάσκεψη της Ρώμης και κατά τη συνάντηση της ομάδας εργασίας ώστε σε όσα θέματα συμφωνούμε αλλά και σε όσα δεν συμφωνούμε να συζητηθούν στη συνομάδα εργασίας πριν από τη Ρώμη. Επανερχόμενος ε, στο πρόγραμμά μας, στην ενότητα αυτή, θα ήθελα να ασχοληθούμε με τον τρόπο αντιμετώπισης των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ένωσης. Η συγκητής του θέματος είναι ο Πιέρ Κάρλο Παντοάν, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, στον οποίο θα μπορέσετε να απευθύνετε τις ερωτήσεις ή τυχόν παρατηρήσεις συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα που έχετε στο φάκελό σας και δίνοντάς σας τη γραμματεία. Με ενημερώνουν ότι ήδη αρκετοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει να λάβουν το λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ακολουθήσουμε την ίδια σειρά όπως και προηγουμένως και τον ίδιο χρόνο. Δηλαδή θα περιοριστούμε στα δύο λεπτά και θα έχουμε τέσσερις ομιλητάς από τα Εθνικά Κοινοβούλια και έναν ομιλητή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Παντουάν, έχετε το λόγο. Πού Where? Where is? Εδώ κάτω κάθεται, ήθελα να κάνει παρουσίαση με το... Α, yes. Okay, okay. Uh, thank you, Mr. Chairman, and... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ βρίσκομαι, δεν με βλέπετε. Θα ανέβω στο βήμα όμως μετά τη σύντομη παρουσίασή μου. Θα ήθελα να θέσω το πλαίσιο των δημοσιονομικών ανισορροπιών στην Ευρώπη με βάση τις προβλέψεις του ΩΣΑ που δημοσιεύθηκαν ε, πριν λίγους μήνες. Το γράφημα αυτό είναι οικείο σε όλους σας, στην παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε, να... Βλέπουμε ανάκαμψη, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες. Έχουμε στα αριστερά τις αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες, τις αναπτυσσόμενες, οι οποίες αναπτύσσονται πιο γρήγορα από ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες και βλέπετε τις χώρες του ευρώ, στις οποίες ε, έχουμε επιτέλους ανάπτυξη περισσότερες από αυτές, αλλά αργή ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι η ε, ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει δυσκολία στην ε, ανάκαμψη στην παραγωγή. Σε προηγούμενες παγκόσμιες υφέσεις ήταν πολύ πιο γρήγορη η ανάκαμψη και με πολύ λιγότερη ζημιά ε, στη δυνατότητα παραγωγής και στην ε, ανεργία, στην απασχόληση. Τα, τα κίνητρα λοιπόν της ανάπτυξης είναι πολύ πιο αδύναμα από ό,τι θα θέλαμε. Καταρχάς, οι επενδύσεις κεφαλογικών αγαθών ε, φαίνονται να είναι χαμηλότερες από ό,τι θα θέλαμε, ε, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Επίσης βλέπουμε ύφεση στις πιστώσεις. Αυτό είναι περισσότερο ευρωπαϊκό πρόβλημα Βλέπουμε ότι αλλού στις Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και σε κάποιο βαθμό στη Ιαπωνία ε, υπάρχει πιο ικανοποιητική πρόοδος. Και επίσης όλοι γνωρίζετε ότι η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει ανεργία, μάλιστα ανεργία στο σύνολο του όσα, ενώ βλέπουμε μείωση της ανεργίας στις Ηνωμένε Πολιτείε και σταθερές χαμηλές τιμές στη Ιαπωνία. Θα ήθελα λοιπόν να φτάσω στο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, τις ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες ε, στην ε, ζώνη του ευρώ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ανισορροπίες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Έχουμε το ισοζύγιο πληρωμών, υπάρχουν όμως ανισορροπίες και στην νομισματική ένωση, τον τρόπο λειτουργίας της, τον, τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, ανισορροπία στον, στην ανταγωνιστικότητα και, και χρειάζονται εδώ προσαρμογές σε διάφορους ε, τομείς, ε, μακροοικονομικές προσαρμογές και διαρθρωτικές. Αυτό εδώ μας θυμίζει αυτά που έχουμε δει στη ζώνη του ευρώ στο παρελθόν. Έχουν λοιπόν αυξηθεί οι ανισορροπία στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών στην, στην ε, ζώνη του ευρώ. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αποκατάσταση των ε, ανισορροπιών. Αλλά γιατί αναπτύχθηκαν αυτές οι ανισορροπίες. Υπάρχουν ε, διάφοροι λόγοι. Πριν την κρίση, όπως θα θυμάστε, η λεγόμενη περιφέρεια τη ζώνη του ευρώ αναπτυσσόταν πολύ περισσότερο από τον πυρήνα της ζώνης του ευρώ. Ενώ τώρα βλέπουμε ακριβώς ε, την αντίθετη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μία, μη, ένα μη βιώσιμο μοτίβο ανάπτυξης, ανισορροπίες στην ανταγωνιστικότητα, ήταν όμως και αποτέλεσμα ανισορροπιών στον μηχανισμό κατανομής πιστώσεων εντός ε, της ζώνης του ευρώ δίδονταν πιστώσεις στην περιφέρεια και είχαμε έτσι ένα μηχανισμό ανάπτυξης μη, βιώσιμος, μη βιώσιμο. Και κατά την αποκατάσταση των ανισορροπιών δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα διαρθωτικά μέτρα από την πρόοδο στην Τραπεζική Ένωση, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη σύνοδο. Αυτό έχει επιδεινωθεί από αυτά που κάνουν οι αγορές και αυτό δεν είναι κάτι νέο. Για πολύ καιρό οι αγορές φαίνονταν να κοιμόντουσαν, δεν υπήρχε αξιολόγηση του κινδύνου για πολύ καιρό μετά τη δημιουργία της ζώνης του ευρώ. Με το ξεκίνημα της κρίσης όμως, μετά το 2009, είδαμε ξαφνικά πολλές αξιολογήσεις κινδύνου άρχισαν να αυξάνονται τα spreads και άρχισαν ε, να μειώνονται πάλι μόνο μετά από πολλή προσπάθεια. Υπάρχει λοιπόν ε, και εδώ ανάγκη διόρθωση διορθωτικών μέτρων. Δυστυχώς ε, τα spread στα κρατικά ομόλογα μας δείχνουν τον κατακαιρματισμό που υπάρχει. Έχουμε το παράδοξο της νομισματικής ένωσης κατακαιρματισμένων νόμων χρηματοπιστωτικών αγορών. Γι' αυτό τα ωφέλη μιας κοινή νομισματικής πολιτικής ε, δεν μοιράζονται ίσα σε όλη την νομισματική ένωση. Αυτό είναι κακό και για την ανάπτυξη και για την αποκατάσταση της ισορροπίας. Θα πρέπει λοιπόν να σημειωθεί πρόοδο στην Τραπεζική Ένωση. Απομένουν πολλά να γίνουν. Πολλά ήδη έχουν γίνει ε, από διαρθρωτικής πλευράς. Το σχέδιο αυτό που βλέπετε βασίζεται σε έναν δίχτυ που χρησιμοποιούμε στον ΩΣΑ για να διαπιστώσουμε την πρόοδο στα, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Βλέπουμε λοιπόν ε, στη ζώνη του ευρώ ότι έχει σημειωθεί πρόοδος πολύ μεγαλύτερη από ότι ε, αυτή που αντιστοιχεί στο μέσο όρο του όσα έχουν γίνει πολλά ήδη δηλαδή. Επίσης έχουν γίνει πολλά στις ε, αγορές εργασίας και στις ε, άλλες αγορές. Ένα πρόβλημα όμως κατά την προσαρμογή στη ζώνη του ευρώ είναι ότι ενώ έχουν επιτευχθεί πολλά όσον αφορά την απασχόληση, την αγορά εργασίας, πρέπει να γίνουν πολλά άλλα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ώστε τα ωφέλη των πιο αποτελεσματικών αγορών ε, να ε, μεταφραστούν σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αυτό αρχίζει να αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που γίνονται οι προσαρμογές. Βλέπετε εδώ την ε, βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε χώρες της περιφέρειας. Σε μεγάλο βαθμό έχει μειωθεί η ζήτηση, έτσι έχουν μειωθεί οι εισαγωγές, αλλά στο... αλλά έχουν ληφθεί μέτρα για να βελτιωθούν οι εξαγωγές. Όλα αυτά όμως ε, είναι άνισα, ασύμετρα. Ε, πολύ λίγη προσαρμογή έχει γίνει σε χώρες ε, πλεονασματικές και έτσι το συνολικό ισοζύγιο της ζώνης του ευρώ παρουσιάζει σε όλο μεγαλύτερο βαθμό πλεόνασμα, κάτι που μπορεί να πιέσει το ευρώ προς τα πάνω, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αποπληθωρισμό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή είναι μια συνολική ανισορροπία η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τέλος, το βασικό ερώτημα μου είναι το εξής. Καλά νέα είναι ότι η ανάπτυξη αυξάνεται ιδιαίτερα στις χώρες της περιφέρειας, ιδιαίτερα λόγω των εξαγωγών. Το θέμα είναι όμως αυτός ο μηχανισμός ανάπτυξης πόσο καιρό μπορεί να επιβιώσει. Η Ευρώπη χρειάζεται βιώσιμη ανάπτυξη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα της ανεργίας των νέων. Αυτό θα αρχίσει να γίνεται όταν δούμε περισσότερες επενδύσεις ώστε τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη από τις ε, εξαγωγές ε, να ε, διοχετευτούν σε επενδύσεις. Θα κλείσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα ανέβω στο βήμα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Αλένα Γκαϊντοσκόβα, πρώτη αντιπρόεδρος της Ρουσίας της Δημοκρατίας.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 Τώρα γενικότερα και εγώ ήθελα να μιλήσω προηγουμένω αλλά δεν μπόρεσα. Πρώτα απ' όλα αρχίζοντα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ελληνική Προεδρία που οργάνωσαν αυτή την διακοινοβουλευτική διάσκεψη. Διότι θεωρώ ότι ο διακοινοβουλευτικός διάλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις Εθνικές Βουλές δεν είναι μόνο κλειδί για τα κράτη-μέλη, αλλά διότι και η ευρωπαϊκή πολιτική γενικότερα δεν μπορεί να επιτύχει εάν δεν ε, μοιραστεί κάποια πράγματα με τις Εθνικές Βουλές. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που οργανώσετε αυτή την διάσκεψη. Πρέπει να πω ότι στην ε, τσεχική δημοκρατία μετά τις τελευταίες εκλογές έχουμε συμμαχία μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και ε, συντηρητικών. Και μέσω της συνεργασίας αυτής θέλουμε να πετύχουμε και ακόμη περισσότερα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε να μπορέσει να γίνει η σωστή δημοσιονομική πολιτική, η σωστή τραπεζική έντοση, αλλά να ληφθεί υπόψη και η κοινωνική πλευρά του όλου Θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο σωστό, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί χωρίς να υπάρχουν προσκόμματα σε κάποιες κοινωνίες. Η Τραπεζική Ένωση είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να έχει σαφείς κανόνες και διατάξεις ώστε να έχουμε υγιή δημοσιονομική πολιτική και τραπεζική πολιτική. Και πρέπει όλοι να ενεργήσουμε από κοινού και να εξασφαλιστεί καλή ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Γι' αυτό την κοινωνική διάσταση μην την ξεχνάτε, διότι νομίζω είναι κάτι το οποίο προς το παρόν ελείπει. Το λόγο έχει ο κύριος Ρισάρ Γιάνγκ από τη Γαλλική Ρουσία Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Euh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμεθα. Το κύριο ερώτημα είναι ποιος είναι τελικά ο δικημενικός στόχος αυτών των ανταλλαγών απόψεων και των διακυλευτικών συναντήσεων. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, διότι μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει σε κάθε ε, κοινωνία. Αλλά εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο πρέπει να λάβουμε υπόψη το θέμα της ε, δημοκρατίας και τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του καθενώνας στα πλαίσια αυτής της διακοινοβουλευτικής διάσκεψης. Δεύτερη παρατήρηση. Για την Τραπεζική Ένωση δεν μπόρεσα να κάνω κάποια παρατήρηση προηγουμένως, χαιρετίζω την μεγάλη και ταχεία πρόοδο που επιτεύχθηκε κυρίως όσον αφορά την εποπτεία. Παραμένουν όμως ακόμη δύο σημαντικά προβλήματα. Το θέμα της εξυγίανσης, το θέμα της ε, ε, δημιουργίας των σχετικών ταμείων και το θέμα της διακυβέρνησης. Πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι τις επικρίσεις που έγιναν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι κι άλλα σε εθνικές βουλές ημερίζονται την άποψη αυτή. Πρέπει να προχωρήσουμε, να καταλήξουμε σε μία συμβαστική λύση, αλλά μία καλή συμβαστική λύση, όχι μια κακιά. Πραγματικά λοιπόν πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε το θέμα αυτό της εξυγίανσης να αποτελέσει μια σημαντική πρόοδο. Τώρα, το συγκεκριμένο θέμα το τωρινό, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Θα ήθελα να προβάλλω μία ιδέα που συζητήθηκε ήδη στην Γερουσία, στη Γαλλία, που είναι να δοθεί στην Ευρωζώνη μία ίδια δημοσιονομική αρμοδιότητα ώστε να ενεργεί αντικυκλικά, δηλαδή θετικά σε περίοδους ανάπτυξης και σε θέματα ε, δυσκολιών να μπορεί να κάνει κάτι για τις δαπάνες. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να αποτελέσει ένα από τα μελλοντικά θέματα συζήτηση μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. Αντρέι Χούνκο από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ähm, ähm, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να διευκρινίσω ότι εγώ δεν εκφράζω την άποψη της πλειοψηφίας ε, του Γερμανικού Κοινοβουλίου αλλά της ε, αντιπολίτευσης ε, των Λίνκε. Και στη Γερμανία γίνονται πάρα πολλές αναλύσεις και συζητήσεις γενικά για την ευρωκρίση και για το πρόβλημα των μακροοικονομικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Προηγουμένως, τα γραφήματα που είδαμε, ε, είδαμε ότι η Γερμανία έχει ένα πολύ μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα, πάνω από 6% και με τον τρόπο αυτό ε, είναι και αυτή ένα πρόβλημα στον ε, ευρωχώρο. Γιατί είναι σαφές ότι το πλεόνασμα του ενός κράτους είναι κατ' ουσίαν το έλλειμμα ενός άλλου. Οι ερωτήσεις μου προς τον κύριο Πάντουαν είναι οι εξής. Εσείς συγκεκριμένα τι μέτρα έχετε να προτείνετε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές οι ανισορροπίες. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε εναρμόνιση στο χώρο της Ευρωζώνης αλλά και σε διεθνές επίπεδο θα έλεγα γιατί βλέπουμε ότι προκύπτει σε γενικές γραμμές όλο και μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη τώρα, σε σχέση με αυτά που είπατε. Μιλήσατε για κατακαιρματισμό κατακαιρματισμένο χώρο δανειοδότησης ε, στην Ευρωζώνη. Και είδαμε στα γραφήματα τις εξελίξεις των επιτοκίων από το 2000 μέχρι το 2008 στις διάφορες χώρες της ε, Ευρωζώνης. Είδαμε τα επιτόκια εκείνη την περίοδο εξελίσσονται αρμονικά. Μετά όμως προέκυψε πολύ μεγάλο άνοιγμα της αλυσίδα μέχρι και 14% νομίζω έφτασε το ποσοστό στην Ελλάδα. Άρα δηλαδή εδώ έχω τη δεύτερη μου ερώτηση πώς μπορούμε να ε, καταλήξουμε και σε εναρμόνιση στην Ευρώπη. Επίσης, ε, στο συνάδελφό σας κύριο Γκουρία, το είπα ήδη στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό ότι ο ΑΣΑ χρησιμοποιεί τους όρους ε, συνεργασία και ανάπτυξη. Ίσως σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο μέλλον να χρειαζόμαστε περισσότερο ανάπτυξη από λιτότητα και συνεργασία από ανταγωνιστικότητα. Το λόγο έχει η κυρία Ελιζάμπετ Κιγκού, Πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών της Γαλλικής Εθνοσκυνέλευσης. Ε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παρέμβασή μου αφορά κυρίως την οργάνωση της διακοινοβουλευτικής διάσκεψης. Μία παρατήρηση για την διακυβέρνηση της Ευρωζώνης που προχώρησε τα τελευταίους μήνες με μία σειρά πρωτοβουλειών και αναφέρω την Τραπεζική Ένωση, βλέπουμε ότι η ναι, βγήκε από τις μεγάλες διαταράξεις. Πολλές χώρες ε, έχουν πρόβλημα, αλλά έκαναν πολλά πράγματα και πρέπει να δούμε ποια είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους. Στους μεν όμως ε, επιβάλλονται μέτρα λιτότητες, υπάρχει μια κάποια διαφάνεια, διαφορετικά μέτρα προτείνονται, άρα μπορούμε να έχουμε επιπτώσεις ευρωεκλογέ. Στα πλαίσια αυτής της διάσκεψης νομίζω ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε πλήρως το ρόλο μας. Πιστεύω ότι η διάσκεψη θα πρέπει να συνεδριάζει στις στιγμές τι πολύ σημαντικές για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ιανουάριος και Οκτώβριος δεν είναι οι πιο σημαντικές στιγμές. Για το Μάρτιο λαμβάνονται οι αποφάσεις για τους οικονομικούς ε, προσανατολισμούς. Τότε κάνει τις προτάσεις η Κομισιόν πριν από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου. Και τότε μπορούν να αποφανθούν για τις γενικές γραμμές των σχεδίων προπολισμού τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κατά την άποψή μου πρόκειται για σημεία κλειδιά και οι επιπτώσεις των δικών μας αποφάσεων θα μπορούν να είναι σημαντικές, όσο και στις δικές μας χώρες, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διάσκεψη βεβαίως και θα πρέπει να συνεδριάσει τον Οκτώβριο μετά από τις νομοδοτήσεις των Εθνικών Βουλών. Τώρα, όσον αφορά την διακυβέρνηση, θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμπεράσματα στη διάσκεψη για να δουν τι κάνουμε και οι πολίτες και να καταλήξουν συμπεράσματα με την ε, αρχή της συνένεσης ή με την ενισχυμένη πλειοψηφία όπως την ΚΟΖΑΚ, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, ρυθμίσουμε και τα θέματα αριθμού βουλευτών κτλ. Και η τελευταία μου παρατήρηση αφορά μία, τη σύσταση μιας ειδική επιτροπής που πρέπει να συστήσουμε για τα προβλήματα των χωρών της Ευρωζώνης που θα συζητήσει όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν στην Ευρωζώνη. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι μετά τις ευρωεκλογέ θα πρέπει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συσταθεί μια ειδική τέτοια επιτροπή ή υποεπιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ελίζα Φερέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Um, Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα στους συναδέλφους των Εθνικών Βουλών. Πιστεύω ότι στην Τραπεζική Ένωση πρέπει να προοδεύσουμε αλλά όχι πρόοδο με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, με κάτι το λογικό τουλάχιστον να εγγυηθούμε την αποδοτικότητα στην διαχείριση των προβληματικών τραπεζών, ίση μεταχείριση για οποιαδήποτε τράπεζα, όπου και να βρίσκεται, σε οποιαδήποτε χώρα και θα πρέπει να μην αφήνουμε ε, τους ε, πολίτες και τους καταθέτες στην ε, άκρη των αποφασεών μας. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε και με ποιο μηχανισμό το Συμβούλιο θα μπορέσει να ελέγξει τις θέσεις των κρατών μελών όταν ε, παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τα σημαντικά στοιχεία τα οποία μας παρουσιάσατε για αυτά τα ειδικά θέματα. Βεβαίως, είναι αληθές ότι οι ανισορροπίες οι εμπορικές και των συναλλαγών αυξήθηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πιο λεπτομεριακά τους λόγους για τους οποίες η παγκοσμιοποίηση, η ενιαία εσωτερική αγορά και το κοινωνικό ε, νόμισμα συμπεριφέρθηκαν όπως συμπεριφέρθηκαν. Πρόκειται για δυναμία κάποιων κρατών μελών. Δεύτερον, πιστεύετε ότι στο μέλλον αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα ελέγξουμε ή τι λείπει από την Ευρωζώνη ε, για να αντισταθμίσει κάποιος το θέμα των ε, φυσικών σταθεροποιητών που δεν διαθέτουν κάποιες οικονομίες. Επίσης, οι περισσότερες χώρες της προσαρμογής έκαναν τρομερές περικοπές στα κονδύλια τεχνολογίας και έρευνας ή οτιδήποτε θα τους επέτρεψε να προχωρήσουν στην σύγχρονη κοινωνία σήμερα. Τι έχετε να πείτε ο Φίλιππος Αγενίδης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της ΕΕ, από την Ελλάδα. Ε, ευχαριστώ. Ε, θέλω να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελληνικό Κοινοβούλιο για την επιτυχημένη αυτή συνδιοργάνωση. Οι χώρες σε πρόγραμμα όπως η Ελλάδα καλούνται να μειώσουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα για να θέσουν σε έλεγχο το χρέος. Ταυτόχρονα καλούνται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της εσωτερικής υποτίμησης για να εξουδετερώσουν τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Τον τελευταίο χρόνο παρατηρούμε το εξής παράδοξο στην Ελλάδα. Η χώρα έχει για πρώτη φορά από μετά τον πόλεμο, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά χειροτερεύοντας τη δυναμική του χρέους διότι παρά το γεγονός ότι πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεόνασμα μειώνεται το ονομαστικό ΑΕΠ. Αν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συνεχίσει να στηρίζεται στον αποπληθωρισμό, τότε η δυναμική του χρέους θα χειροτερέψει ενώ δημοσιονομικά ακολουθούμε τη σωστή πολιτική. Για να το αποφύγει αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να έχει όχι αποπληθωρισμό αλλά πληθωρισμό χαμηλότερο από το μέσο όρο των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρατά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη κοντά στο 1% ενώ μπορεί να τον έχει πολύ κοντά στο 2%. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι χώρες με πλεόνασμα πρέπει να έχουν λίγο υψηλότερο πληθωρισμό από τον τρέχοντα για να βοηθήσουν τις χώρες με έλλειμμα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, τον κύριο Πιερ Κάλλο Παντουάν. Έχουν μαζευτεί αρκετές ερωτήσεις για να απαντήσετε. Thank you for all these questions. Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις αυτές. Ελπίζω να σημείωσα σωστά τη σειρά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και συνοπτικά σε κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς να αναφερθώ στο θέμα των ανισορροπιών στην Ευρωζώνη και το τι μπορεί να γίνει, ώστε οι πλεονασματικές χώρες να μετριάσουν τις ανισορροπίες. Υπάρχει μία λύση που θα ωφελήσει και την Ευρωζώνη και την χώρα αυτή καθ' αυτή. πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών ε, σημαίνει λίγες επενδύσεις σε σχέση με τις αποταμιεύσεις. Η σύσταση λοιπόν που δίνει ο ΣΑ πάντα στις πλεονασματικές χώρες στην Ευρωζώνη και αλλού είναι να προωθήσουν τις επενδύσεις, κάτι που μπορεί να γίνει προς όφελος της χώρας, απελευθερώνοντας κάποιους τομείς υπηρεσιών, ακόμα και σε χώρες σαν τη Γερμανία, όπου είναι πολύ ανταγωνιστικός ο τομέας παραγωγής, ο τομέας κατασκευών. Βελτίωση της παραγωγικότητας μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση των υπηρεσιών, κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση των ε, επενδύσεων. Αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη και στη Γερμανία και αλλού, γιατί θα κερδίσουν όλοι. Να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, με τη σειρά που τέθηκαν. Κατακαιρματισμός ε, των πιστώσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Απαιτεί δράση σε διάφορα επίπεδα. Καταρχάς, απαιτεί η σχέση τραπεζών και δημοσίου χρέους ε, να ε, την ή να σταματήσει τελείως. Το δημόσιο χρέος ε, μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αναταράξεων και αυτό οδηγεί σε συνέπειες στους λογαριασμούς των τραπεζών. Θέλουμε όμως να βελτιωθεί και η ανταγωνιστικότητα στις χώρες, ώστε οι τράπεζες ε, να δανείζουν σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Υπάρχει λοιπόν σχέση, υπάρχει συνέργεια ανάμεσα στην πρόοδο στην Τραπεζική Ένωση, τις ε, ε, τα διαφορετικά μέτρα και τα μέτρα προσαρμογής. Και αυτό με οδηγεί στο ερώτημα. Γιατί δεν είδαμε αυτές τις ανισορροπίες πριν την κρίση. Θα θυμάστε όλοι τη συζήτηση στην Ευρώπη σχετικά με το πώς θα οικοτομηθεί η νομισματική ένωση. Και αναφέρθηκαν κυρίως ε, η δημοσιονομική προσαρμογή και η σύγκληση όσον αφορά τον πληθωρισμό. Η κρίση όμως μας θυμίζει ότι οι ανισορροπίες δημιουργούνται εντός της νομισματικής ένωσης, σε κάτι που οδηγεί σε μη βιώσιμες ανισορροπίες και μάλιστα δύο αρνητικούς ε, παράγοντες που προσπάθησα να παρουσιάσω στις ε, διαφάνειές μου. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητα δεν αντιμετωπίζεται σε κάποιε χώρε, επειδή ούτω ή άλλω συνεχίζεται η ανάπτυξη. Αυτό το είδαμε σε πολλέ χώρε τη περιφέρεια. Και η ανάπτυξη συνεχίζεται διότι χρηματοδοτείται με κεφάλαια και επιστώσει που προέρχονται από τις πλεονασματικές χώρες. Έτσι λοιπόν και οι δύο πλευρές ε, ε, φταίνε για τη δημιουργία των ανισορροπιών. Τι θα πρέπει λοιπόν να γίνει. Θα πρέπει να εξαλειφθούν οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα με διαφορετικά μέτρα. Θα πρέπει όμως επίσης να υπάρχει ένα σύστημα πίστοσης που να κατανέμει σωστά τα χρήματα. Έτσι να αποφεύγονται οι φούσκες πιστώσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει και η ζώνη του ευρώ αλλά και άλλες χώρες. Υπάρχουν διάφορα μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν. Υπάρχει η Τραπεζική Ένωση, υπάρχουν όμως ε, και ε, μέτρα προληπτικής εποπτείας, μακροπρόθεσμης προληπτικής εποπτείας. Υπάρχουν λοιπόν πολλά μέσα τα οποία μπορούν να μας, να μας οδηγήσουν σε ένα σύστημα πιστώσεων το οποίο να λειτουργεί σωστά και να κατανέμει σωστά τους πόρους στους τομείς που είναι βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια ανισορροπία που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ζώνη του ευρώ. Πώ μπορούμε να κάνουμε οι ανισορροπίε αυτέ να είναι πιο βιώσιμε, όχι να τι εξαλείψουμε. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα μειώσει το γενικό πλεόνασμα, το οποίο έχει αποπληθωριστικό αποτέλεσμα στην Ευρωζώνη. Αυτό θα αποτελέσει αποτέλεσμα των πολιτικών ανάπτυξης και καλύτερων μηχανισμών κατανομής. Επίσης ρωτήθηκα τι εννοώ όταν λέω διαρθρωτικά μέτρα. Να σας θυμίσω κάτι πολύ γνωστό. Οι περισσότερες προσπάθειες και οι δαπάνες προσαρμογής ιδιαίτερα στην περιφέρεια ήταν αποτέλεσμα δημοσιονομικής εξυγίανση ε, παρά διαρθρωτικών μέτρων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Εγώ σκέφτομαι ιδιαίτερε προσαρμογέ ε, στι αγορέ εργασία, ώστε να υπάρχει καλύτερη ανακατονομή του εργατικού δυναμικού, καλύτερη κατάρτιση των ανθρώπων και καλύτερη στήριξη κατά τη ε, μετάβαση από τη μία θέση εργασία σε κάποια άλλη. Επίσης πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας ώστε το χαμηλότερο κόστος εργασίας να, μεταφερθεί, να μετατραπεί σε χαμηλότερο κόστος για τα προϊόντα. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα σε όλες τις χώρες της περιφέρειας. Θα πρέπει λοιπόν τα διαφορετικά μέτρα να είναι συνολικά ώστε τα ωφέλη από τον έναν τομέα να οδηγούν σε ωφέλη σε άλλους τομείς. Επίσης, ε, να αναφερθώ σε ένα στοιχείο που έχουμε δει στις μεταρρυθμιστικές πολιτικές σε όλο τον κόσμο. Οι διαρθρωτικές ε, αλλαγές έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα ανάμεσα με τη φάση του κύκλου στην οποία βρισκόμαστε. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για να εμφανιστούν τα ωφέλη ή λιγότερος. Θα πρέπει λοιπόν να ε, φροντίσουμε οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις να γίνουν και την κατάλληλη χρονική στιγμή. Συμφωνώ επίσης ότι ο αποπληθωρισμός σε χώρες με υψηλό χρέος είναι πρόβλημα. Μπορεί να είναι ε, καταστροφικό αυτό. Βλέπουμε νομισματική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ γενικά θετική εξέλιξη τιμών ακόμα και στις χώρες που θα πρέπει να αποκαταστήσουν την ισορροπία στις τιμές τους. Είναι αριθμητική, απλή αριθμητική. Εάν πέσουν οι τιμές, εάν πέσει το ονομαστικό ΑΕΠ, τότε δυσκολεύει η προσαρμογή, δεν γίνεται πιο εύκολη. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία και συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε. Αυτό βέβαια απαιτεί προσπάθειες σε επίπεδο ζώνης του ευρώ. Θα πρέπει να δούμε τη δυναμική των τιμών. Απαιτούνται και προσπάθειες σε επίπεδο χώρας για την προσαρμογή των τιμών. Θα πρέπει να γίνει συντονισμό όμως, διότι μόνο ένα κομμάτι της συνολικής αυτής στρατηγικής δεν θα λειτουργήσει. And now? Yes. Say thank you to him. Okay. Thank you, Wir hatten vereinbart, meine, do you have? Okay, please continue. Apologies for that. I forgot to. Κοιτάξτε, ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέχασα να σχολιάσω το θέμα των αυτόματων σταθεροποιητών. Και νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο στην Ευρωζώνη ε, έτσι ώστε με κάποιους ε, μηχανισμούς ε, να βρούμε ένα είδος ε, εξομάλυνσης του κύκλου. Και αυτά αφορά δύο θέματα. Πρώτον, πώς μπορεί κανείς να βρει αυτό, αυτή τη δεξαμηνή πόρων. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή το απαραίτητο και κατάλληλο οργανείο είναι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Αλλά μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Και το άλλο θέμα είναι ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόσουμε έτσι ώστε από αυτή την κοινή δεξαμενή να διοχετεύουμε κονδύλια στις χώρες που τα χρειάζονται. Αυτό μέχρι κάποιο σημείο είναι τεχνικής φύσεως πρόβλημα. Ε, μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν οι ε, πόροι για αγορές, ε, για πολιτικές στην αγορά εργασίας, τους αυτόματους σταθεροποιητές, όλα αυτά είναι μια μακρά συζήτηση και για να εξοικονομούμε χρόνο ε, θέλω να πω ότι συμφωνώ επί της αρχής. Η ε, Οικονομική και Ένωση θα επωφελεί το αν υπήρχε ένας τέτοιος μηχανισμός. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμφωνήσαμε το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη συζήτηση να τη μοιραστούμε το πρώτο ήμιση προείδρευσε ο κύριος Τραγάκης και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τραγάκη και τώρα προεδρεύω εγώ. Έχουμε άλλες ε, έξι ερωτήσεις μέχρι να φτάσουμε στο δεύτερο γύρο των απαντήσεων και δίνω το λόγο στον κύριο Σόρντ από την Εστονία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Αυτό το οποίο όμως είναι σαφές είναι ότι ο συντονισμός των προϋπολογισμών των κρατών μιλών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συντονιστεί μεταξύ μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πραγματικά να εντείνει ακόμη και το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό. Διαφορετικά θα μπορούσαν οι ανισορροπίες να μεγαλώσουν. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό όμως να πούμε είναι ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός επίσης θα έχει, πρέπει να έχει έναν προσανατολισμό προς την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων. Τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών πρέπει να πω ότι καταβάλαμε προσπάθειες που απέδωσαν. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, να ενθαρρύνουμε την ε, μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς και όσον αφορά τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις συνθήκες που θα μας βοηθήσουν. Έχει αρχίσει η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, έχουν τεθεί κάποιες προτεραιότητες και οι συστάσεις που έχουν γίνει θα πρέπει να πάρουν σάρκα και ωστά, να γίνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Διότι σε πολλές περιπτώσεις υπογράφονται συμφωνίες αλλά θα πρέπει να τεθούν και σε εφαρμογή ώστε να έχουμε αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Επίσης, δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε την αγορά εργασίας και τον ανταγωνισμό που υπάρχει. Στην ε, Εστονία θελήσαμε να αυξήσουμε την παραγωγή γιατί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και το σύστημα παιδείας επίσης πρέπει να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε στις σημερινές ανάγκες. Η οικονομία μας στην Εστονία πρέπει να πω ότι επίσης ε, ε, στην αρχή της ε, κρίσης αντιμετώπισε πρόβλημα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε εξυγίανση, να δημιουργήσουμε αποθεματικό και πιστεύω ότι η διάσκεψή μας είναι πραγματικά μια προστιθέμενη αξία που μας επιτρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τις οικονομικές πολιτικές μας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Um, um, Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλώ ε, στο όνομα των χριστιανοδημοκρατών ε, των κάτω χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ακριβή περιγραφή των θεμάτων που έχουμε εδώ πέρα. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μας είχατε μοιράσει τις διαφάνειες ε, πριν την ομιλία σας, ώστε να διαφρόσουμε καλύτερα τη συζήτηση. Θα συμφωνήσω με τους ε, τρεις προλαλήσαντες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια μικρή επιτροπή που θα συζητήσει την ε, οργάνωση όλης αυτής της συνέλευσης ε, για την επόμενη φορά. Ακούμε διάφορες ιδέες, μια μεταρρυθμιστική συνθήκη, ε, προϋπολογισμός ε, της ζώνης του ευρώ κλπ. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να διαρθρωθεί, να διαρθρωθεί η συζήτηση τη στιγμή που συμμετέχουν 28 κράτη-μέλη. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που θα ήθελα να θέσω στον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Πολύ ευχαρίστω θα το συζητήσω και κατηδίαν μαζί του. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση. Ακούω να λένε ότι πρέπει να ε, σπάσει η σύνδεση ανάμεσα στις ε, τράπεζες και το δημόσιο χρέος. Είδαμε την Ιρλανδία να καταραίει λόγω μιας τράπεζας. Και εάν έχουμε ακόμα περισσότερες συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ευρώπη, θα μπορέσουν να ε, ανατρέψουν όλο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν να φροντίσουμε να μην έχουμε υπερβολικά μεγάλες τράπεζες. Θα ήθελα να ακούσω τη θέση του ΩΣΑ για τις τράπεζες. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Χάνκο. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα σχετικά με τις προτάσεις του ΩΣΑ ώστε να διασφαλιστεί οι πλεονασματικές χώρες όπως είναι οι κάτω χώρες τι είδους μέτρα προτείνει για τις ε, πλεονασματικές αυτές χώρες. Ευχαριστώ κύριο Σόρση Σίκεν. He's not here. So, Mr. Okay, δεν είναι εδώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που οργανώσατε αυτή τη συνάντηση που γίνεται την κατάλληλη στιγμή. Κάποιες παρατηρήσεις που ίσως σας φαρούν εκτός θέματος, γιατί ήθελα στην αρχή της Ολομελίας να λάβω το λόγο. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις τρεις ε, επιτροπές σήμερα το απόγευμα, της ε, απασχόλησης, του προπολογισμού και της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Θα ήθελα να προτείνω και την ε, συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Ξέρουμε ότι σε κάθε δημοκρατία τα κοινοβούλια ελέγχουν και την εκτελεστική εξουσία αλλά και τα του προπολογισμού. Εμείς αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να ασκήσουμε έλεγχο προπολογισμού και πολιτικό έλεγχο πλήρως μόνο με έναν εξωτερικό οικονομικό ελεγκτή ε, κάνουμε τη δουλειά μας και πολλοί ενοχλούνται από αυτόν τον ε, μηχανισμό που είναι μια εταιρεία ε, με έδρα το Λουξεμβούργο που κάνει το ελέγχου αυτού. Εφόσον μιλούμε λοιπόν για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Από όσον ξέρω, οι χώρες εκτός Ευρωζώνης συνεδριάζουν διαφορετικά από εμείς. Και εγώ ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση κύριο Βαν Μιλούμε πολύ για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Πώς οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα εφαρμόσουν τη διάταξη της συνθήκης την οποία θα πρέπει, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ευρωεκλογέ για να κάνουν κάποια πρόταση για τον ορισμό του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πρωταρχή σημασία στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι γίνονται κάποιες συμφωνίες εκτός ε, εκλογέων. Ξέρουμε ότι εμείς ε, πριν από τις εκλογές πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι προτάσεις που θα κάνουν τις, ε, ε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Θα ήθελα να μου πει ο κύριος Βαν τι έχουν κατά νου οι κρατών και ε, κυβερνήσεων. Επίσης, προβλέπεται στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 μια ρήτρα που λέγει ότι θα πρέπει να λειτουργεί σωστά και με αυτόν τον τρόπο η δημοκρατία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας το έλεγα αυτό, θα σας το έλεγα αυτό στο τέλος της συνεδρίας, αλλά η τελευταία ερώτηση δεν έχει καμία σχέση με το άρθρο 13. Εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Πάολο Κουέρ. Ναι. Συμφωνώ σχετικά με την ε, οικονομική εικόνα που σχεδιάσατε, που σκιαγραφίσατε. Στην Ευρωζώνη είχαμε δύο ε, υφέσεις ε, τα τελευταία χρόνια και τώρα πλέον η Ευρωζώνη μοιάζει να ανακάμπτει. Πολύ μικρή ανάκαμψη της τάξης του 1% και γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν με τον τρόπο αυτό να επιληθούν σημαντικά προβλήματα σε πολλές ε, χώρες μέλη προηγούμενη μας ε, πριν από λίγο ακούσαμε ότι ε, θα μπορούσαν να θεωρηθεί ότι τα προγράμματα λιτότητας έχουν θετικά αποτέλεσμα. Άρα δηλαδή για να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα, ανάπτυξη, απλά χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη, πιο ευέλικτη εφαρμογή. Αυτά ακούσαμε. Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες όσον αφορά αυτές τις προβλέψεις, γιατί αν δείτε λιγάκι τι θα γίνει στο μέλλον, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η λιτότητα θα περιοριστεί λόγω της νέας ευέλικτης προσέγγισης των Βρυξελών, νομίζω ότι αυτή η προσαρμογή δεν θα μπορέσει να επιλύσει τα σημαντικά προβλήματα της Ευρωζώνης, κυρίως των περιφερειακών κρατών. Επιπλέον, η εσωτερική υποτίμηση στην οποία αναφερθήκατε, δηλαδή η περικοπή των μισθών και των τιμών ε, σε όλες σχεδόν τις χώρες, προφανώς και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους και τις εξαγωγές. Αλλά η Ευρωζώνη στο σύνολό της ε, θα αναγκαστεί να ακολουθήσει ένα μοντέλο αύξησης των εξαγωγών. Η πιο πλούσια χώρα της Ευρωζώνης θα εξαρτάται απόλυτα από τους ε, Κινέζους καταναλωτές, τους Ταϊλανδούς, ε, όλους αυτούς. Έτσι λοιπόν κάτω από αυτό το πρίσμα, κατά την άποψή μας, ε, πρέπει να φοβόμαστε ότι με αυτές τις πολιτικές δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη, αλλά θα αντιμετωπίσουμε στασιμότητα στο μέλλον. Αυτή θα είναι η τάση. Πρόσφατα η Γενική Διεθνής Αρμόδια για τα Οικονομικά Θέματα δημοσίευσε μια έκθεση που δείχνει ότι αν τα επόμενα 10 χρόνια δεν αλλάξει κάτι, το ε, κατακεφαλή ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά το μέγιστο 1% και ε, το κατακεφαλή ε, ΑΕΠ θα μειωθεί θα επανέλθει στο 1965 περίπου. Έτσι λοιπόν η δική μου η ερώτηση είναι η εξής. Σίγουρα οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές, αλλά η μακροοικονομική πολιτική σε επίπεδο ευρωζώνης είναι πολύ πιο σημαντική, όσο σημαντικές και αν είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η μακροοικονομική πολιτική δεν είναι ουδέτερη. Έτσι λοιπόν, αν συγκρίνουμε σήμερα τις ΗΠΑ Πολιτείες και την Ιαπωνία με την ε, Ευρωζώνη θα διαπιστώσουμε ότι οι μακροοικονομικές διαφορές είναι ο σημαντικότερος λόγος γιατί ε, διαλύεται αυτή η Ευρωζώνη και θα ήθελα να γνωρίζω την άποψή σας επ' αυτού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ε, κύριος Φραντσέσκο Καριέλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα Θέλω να σας ε, επισημάνω το σύμφωνο δημοσιονομικής ε, σταθερότητας κάτω από όμως από νομικό πρίσμα. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω. Να πάμε στην 1η Ιανουαρίου του 1999 όταν ε, πρωτοεισήχθη το ευρώ, το νέο ευρωπαϊκό νόμισμα. Τότε λοιπόν την 1η Ιανουαρίου του 1999 στις αγορές εμφανίστηκε ένα πειθαρχημένο νόμισμα με βάση τις ε, μελέτες που γνωρίζουμε, με μια σχετική συμφωνία που είχε επιτευχθεί. Αυτή όμως η συμφωνία δεν είχε καμία σχέση με την ε, πειθαρχία που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, ο κανονισμός 1466 είναι σε αντίθεση με το άρθρο 104 του συμφώνου. Έτσι λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, σε, αυτή, σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ένας πρώην Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, ο καθηγητής κ. Γκουαρίνο. Και από ό,τι θυμάμαι σήμερα, σε καμία χώρα της Ευρώπης ούτε σε αυτό το κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, κανείς δεν διαφώνησε με αυτή την παραδοχή. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Τουλάχιστον αυτές τις τρεις ε, ημέρες η συνέλευσή μας ας δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή ο κανονισμός 1466 είναι ο ίδιος ή όχι με, το, με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπήρχε την εποχή εκείνη. Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί ο καθηγητής Γκουαρίνο λέει Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον κανονισμό 1466 ε, και πρέπει να πω ότι γίνεται αναφορά στη δέσμευση, στις υποχρεώσεις που προβλέπει ο κανονισμός 1466. Αυτές οι δεσμεύσεις μειώνουν τη δυνατότητα κάθε κράτους να προβεί σε οικονομικούς χειρισμούς. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει αυτός ο σοφός. Αλλά κατά την άποψή μου αυτό το νομικό ερώτημα χρήζει απάντησης από τη συνέλευσή μας. Πρόεδρος, ε, έχω ακόμα ένα μιλητή στον κατάλογό μου. Τον κύριο Οικοαπημένος από τη Λετωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία ειδική ερώτηση για τον κύριο Παντοάν. Εμείς υποφέραμε πολύ, όπως ξέρετε, από την οικονομική κρίση. Η ποιότητα ζωής υποβαθμίστηκε Και αν μου επιτρέψετε θα μιλήσω τη μετρική μου γλώσσα. Πρέπει λοιπόν να σας πω το εξής. Το ΑΕΠ, το δικό μας, είναι το, τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση αυτό της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Και θα χρειαστούμε γενιές ολόκληρες για να μπορέσουμε να είμαστε σε κατάσταση ευημερίας. Έχουμε πολύ χαμηλά επίπεδα όσον αφορά το ΑΕΠ Και περιορισμένη ανάπτυξη. Δεν είναι εύκολο να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές. Και διαρωτώ εάν μπορούμε κάτι για να αυξήσουμε τις πιστώσεις μας, για να τηρήσουμε το δημοσιονομικό σύμφωνο. Αυτό όμω δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει με τη βελτίωση των συνθήκων διαβίβαση των πολιτών. Ποια είναι η αποφάσεις Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις προς τον ομιλητή μας, τον κύριο Παντουμάν. Εάν όχι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις που υποβάλλετε και να δώσω το λόγο στον ομιλητή. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις έτσι όπως τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα, το θέμα της βελτίωσης των ισολογισμών των τραπεζών. Πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία. Ξέρουμε ότι το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή διέρχεται μία διαδικασία ε, αξιολόγησης και ξέρουμε ότι γίνονται και τα περίφημα τεστ αντοχής για τις τράπεζες περιμένουμε να υπάρχει μεγαλύτερη πρόοδος προς την επίτευξη της Τραπεζικής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλα τα τραπεζικά ιδρύματα να λειτουργούν τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να ενισχυθούν οι τράπεζες. Όλη αυτή η διαδικασία, κατά την άποψή μου, είναι πολύ σημαντική και αυτό που συνιστά όσα είναι και τα stress τεστ και όλη η αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των τραπεζών να γίνουν με διαφανή τρόπο. Πράγμα που δεν είχε γίνει στο παρελθόν με αυτόν τον τρόπο, ούτε εδώ ούτε στη ΣΥΠΑ. Όσον αφορά το δίλημα το Ολλανδικό, αν μπορώ να το πω έτσι, πώς μπορούν οι χώρες λοιπόν που έχουν το πλεόνασμα να προχωρήσουν. Η σύσταση της Γερμανίας εδώ είναι χρήσιμη. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να μπορέσει να αφιερωθεί περισσότερο η χώρα στον εσωτερικό ανταγωνισμό και στην βελτίωση των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα με τη λήψη διαφόρων μέτρων, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει και τις προσαρμογές του προϋπολογισμού ώστε να αυξηθούν τα έσοδα. Ο κύριος Γκαριέρη έφεσε το εξή θέμα. Αν θα πρέπει να αφοσιωθούμε μόνο στα θέματα της εξηγήνσης... και να μην κάνουμε τίποτε για την βελτίωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Όχι. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση κάνουμε είναι πιο αδύναμη εάν δεν δούμε και την ε, άμβληση των ε, ε, μακροπρόθεσμων ανισορροπιών. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές και στις διαρθρωτικές μεταβλήσεις. Τώρα, από πού θα μπορούσε να βελτιωθεί στην παρούσα κατάσταση η αύξηση της ζήτησης με οικονομικό. Εγώ δεν έχω το μαγικό ραβδάκι στα χέρια μου, όπως λένε και στη Γαλλία, αλλά θα πρέπει να δούμε προς τα πού θα πρέπει να στραφούμε. Πρώτα απ' όλα, η ε, σφαιρική αν θέλετε η παγκόσμια ζήτηση και καλό είναι το ότι οι αναδυόμενες οικονομίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Πράγμα το οποίο αν θέλετε δίνει μια κάποια όθηση στις δικές μας εξαγωγές αλλά τίποτε δεν είναι από μόνο του επαρκές. Πρέπει να συνδυαστούν διάφορα μέτρα. Η πολιτική της ενιαίας εσωτερικής αγοράς μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Το λέω αυτό μεγαλύτερη πειθό από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Μετά από την ε, εμπειρία της ε, ε, επιθετικής νομεσβήτης πολιτικής των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας μάθαμε κάποια πράγματα από την Κίνα. Μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα και μέσοπρόθεσμα αυτή η επιθετική νομισματική πολιτική σωστή για να μπορέσει η ιδιωτική ε, κατανάλωση να αυξηθεί. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποια μαθήματα από αυτά τα οποία από κάτι το παρεμφερές που έγινε στο θέμα αυτό τη είπα. Επίσης, όσα σε πολλές περιπτώσεις συνιστά να υπάρχουν ε, ευρωπαϊκά προγράμματα επενδυτικά με ομόλογα ανάλογα με τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης βάσει κάποιων μέσα Επίσης, τι μπορούμε να κάνουμε με τη δημοσιονομική πολιτική σήμερα στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων. Κατά την άποψή μου, μπορούμε να κάνουμε σε δύο τομείς πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα με την ταχύτητα με την οποία προχωρεί η δημοσιονομική εξυγίανση και σήμερα βλέπουμε ότι ε, ο λόγος όσον αφορά το θέμα αυτό μειώνεται σε σχέση με το προηγούμενο και δεύτερον όπως αποδεικνύεται, βλέπουμε ότι για κάποια ε, έσοδα θα πρέπει να αλλάξουμε την ε, σύνδεση, την σύνθεση του συνόλου των κονδυλίων που τα απαρτίζουν. Ίσως αυτά είναι περιθωριακά θέματα, αλλά επιμέρους. Ε, αλλά αν τα προσθέσετε σίγουρα μπορείτε να δημιουργήσετε μία δυναμική στην ζήτηση στην Ευρώπη και τελειώνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα τελευταία 10 με 15 χρόνια δυνητικά η ανάπτυξη μειώθηκε. Καλό είναι να έχουμε λοιπόν ε, ε, ε, μέτρα τα οποία θα μας βοηθήσουν ε, βραχυπρόθεσμα στην ανάπτυξη, αλλά και το μικροπρόθεσμα δεν θα πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Ξέχασα το ερώτημα της λεπτομέρειες παρά το γεγονός ότι δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτησή σας. Είπατε εσείς μπορούμε να ε, συνδυάσουμε το δημοσιονομικό σύμφωνο με την ανάπτυξη. Ναι, απαντώ, για τους λόγους που προανέφερα. Και διότι, εάν δεν... Εάν υπάρχει η κατάλληλη ε, ε, δυναμική στην αγορά μπορούν, ε, μπορεί ο δανεισμός να μειωθεί άρα να προχωρήσει η οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Πέρα από το πρόγραμμα του άρθρου 13 και προς ενημέρωση όλων, θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα του Σοπεωτή που απίφθινε προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου και που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε πολύ σαφή διαδικασία όσον αφορά τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι πολιτικές ομάδες δεσμεύθηκαν πριν τις ευρωεκλογέ να παρουσιάσουν τον υποψήφιό τους ή την υποψήφιά τους ε, για πρόεδρο του, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, οι σοσιαλδημοκράτες το έκαναν ήδη. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στους φιλελεύθερους ισοψηφούν όλοι Λιρέν και ο Γκίχε Φερχόφστατ. Οι πράσινοι διεξάγουν επιγραμμικά μια εσωτερική ψηφοφορία. Και στο ΕΛΚ ε, θα ληφθεί απόφαση 6-7 Μαρτίου στο Δουβλίνο μεταξύ διαφόρων υποψηφίων. Πριν τις ευρωεκλογές λοιπόν θα παρουσιάσουν τον υποψήφιό τους για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπτωση που έχουν την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν αδύνατο, ανέθυνο θα ήταν αν το Συμβούλιο ήδη τώρα έλεγε κάτι. Το Ευρωκοινοβούλιο εμέσως ορίζει τον πρόεδρο της Επιτροπής. Τα ονόματα είναι γνωστά πριν τις ευρωεκλογέ. Έτσι λοιπόν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο αποτέλεσμα των εκλογών και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε υποψήφιος όμως πρέπει να συγκεντρώσει ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Η διαδικασία αυτή λοιπόν θα είναι ένας ε, συμβιβασμός που θα εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εκλογών, από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Οι ψηφοφόροι όμως ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν τόση επιρροή, δεν είχαν τόσες πληροφορίες εκ των προτέρων. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πάντως ε, χρειάζονται πλειοψηφία δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η ερώτηση τέθηκε σε έναν απόντα και δεν είχε σχέση με το θέμα της διάσκεψης αυτής. Επί παρεξήγηση. Ξέρω ότι στην αίθουσα αυτή υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Θα πρέπει να επανέλθουμε στην ουσία της διάσκεψης αυτής. Είπαμε, είπε και ο Αντιπρόεδρος κ. Τραγάκης, ότι μετά την διάσκεψη αυτή θα ξεκινήσει μια διαδικασία με βάση τα υπάρχοντα έγγραφα και τις τροπολογίες. Θα υπάρξει μια ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με το θέμα της διαδικασίας. το προσεχές διήμερο λοιπόν θα ήθελα να ασχοληθούμε με την ουσία και όχι με το τυπικό. Η διάσκεψη αυτή έχει τη βάση της στο άρθρο 13. Η διάσκεψη αυτή είναι ευρύτερη όσον αφορά τα θέματα που συζητάμε από οποιαδήποτε άλλη, διότι συνδέσαμε το άρθρο 13 με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τις δυόμιση αυτές μέρες. Το άρθρο 13 είναι βάση της διάσκεψης αυτής και έχει ως θέμα το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Δεν πρόκειται για διάσκεψη ΚΟΣΑΚ. Έχει τη βάση της στο άρθρο 13 στις αποφάσεις της Λευκοσίας και στόχο έχει μια δημοκρατική, διαφανή ανταλλαγή απόψεων πάνω στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Και γι' αυτό έχουμε συγκεντρωθεί εδώ. διότι στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν, με, δεν ασχολείται με τα θέματα αυτά μόνο μία επιτροπή. Είναι θέματα Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Απασχόλησης, της ε, Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπάρχουν και άλλες επιτροπές. Και θελήσαμε στη συζήτηση αυτή να συμμετέχουν όλες οι επιτροπές αυτές. Είναι δύσκολο όμως να ρυθμιστεί αυτό. διότι ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ζητάνε η Επιτροπή Προϋπολογισμού, η Επιτροπή Απασχόλησης, η Κοινωνική Επιτροπή να συμμετέχουν στη σχετική συζήτηση. Πόσο μάλλον λοιπόν με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε την Τετάρτη πώς θα το οργανώσουμε. Υπάρχουν πάντα διαφορετικές απόψεις. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες. Γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε απλά να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και να εξάγουμε συμπεράσματα από τις εμπειρίες των άλλων και από τον διάλογο. Παρακαλώ λοιπόν να επιδείξετε κατανόηση. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βρίσκονται υπό εξέλιξη. Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν οι Γενικοί Γραμματείς των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συζητήσουν πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία, πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλα όμως όσα γίνονται θα ληφθούν υπόψη και στην επόμενη συνάντηση στη Ρώμη. Και αυτά που που συζητήσαμε στο Βίλνιους. Επιθυμία μας είναι λοιπόν να συνεχίσουμε τις εργασίες αυτές. Δεν θέλουμε όμως να χαθούμε στις λεπτομέρειες, διότι έτσι δεν θα φτάσουμε ποτέ στη συζήτηση επί της ουσίας. Το θέμα λοιπόν είναι να μην συζητάμε ποιος θα με πόσους από ποια επιτροπή, Θέλουμε να εργαστούμε με συνενετικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε επί της ουσίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις σας. Οι πολιτικές ομάδες έχουν τώρα γεύμα και συνάντηση και αύριο το πρωί θα ξανασυναντηθούμε στις 9.30 και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση σχετικά με τις δραστηριότητες των κοινοβουλίων και την Τρόικα. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί.